Κυρίες και κύριοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού και Μεταφορών. Έχουμε καταρχήν την ημέρη διάταξη. Έχω μία μάλλον θλιβερή ανακοίνωση να σας κάνω. διότι η κυρία Ουρίκε Μπάρτλιτ Λάρσεν που ήταν η αναπληρωτής πρεσβευτής από τη σουηδική πλευρά και μέλος της μόνιμης ε, αντιπροσωπείας από τη σουηδική πλευρά μας άφησε στις 5 Νοεμβρίου, νομίζω ότι έπασε από καρκίνο. Με την ε, άδειά σας λοιπόν, θα ήθελα να αποστείλω μια επιστολή προς τον Υπουργό Μεταφορών της Σουηδίας, εξ ονόματος Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας για τον θάνατο της κυρίας Λάσεν. Και θα θέλαμε να ζητήσουμε τα συλληπιτήρια αυτά να διαβιβαστούν στους οικείους και στους φίλους της. Εάν συμφωνείτε λοιπόν, θα το πράξω αυτό ήδη την, μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Σύμφωνοι. Ευχαριστώ. Στα θέματα τώρα της ημερήσιας διάταξης, έχουμε καταρχήν την έγκριση της ημερήσιας διάταξης που είναι ενώπιόν σας. Έχετε σχόλια. Εάν όχι, μπορώ να θεωρήσω ότι έχετε εγκρίνει την ημερησία διάταξη αυτή τη συνεδρίαση. Στη συνέχεια, έχουμε την έγκριση των πρακτικών. Τη 5 η και 6ης Οκτωβρίου μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά. Σας ευχαριστώ. Το επόμενο σημείο είναι η ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σε σχέση με την εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και κυρία Χούτμαν που είναι υπεύθυνη για τα θέματα αυτά θα λάβει το λόγο εξ της Κομισιόν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, η Κομισιόν έχει εγγύψει στα θέματα των δικαιωμάτων των επιβατών των αεροπορικών συγκοινωνιών με ιδιαίτερα ενδελεχή τρόπο πρόσφατα. Γνωρίζουμε ότι ο τομέας αυτός έχει παίξει ένα πρωτοπόρο ρόλο στο άνοιγμα των αγορών Έχουμε πάνω από 400 εταιρείε οι οποίες ασκούν αεροπορικέ μεταφορές και περίπου 700, 750, εκατομμύρια επιβατών ετησίω μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πεπισμένοι λοιπόν ότι οι βελτιώσει στον τομέα αυτό θα ανοίξουν το δρόμο και για άλλου τρόπου μεταφορών. Όπως ξέρετε, από το Δεκέμβριο θα τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός για τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών. Ε, Επίση, έχει εγκρίνει το Συμβούλιο ένα αντίστοιχο κανονισμό για τις θαλάσσιες μεταφορές και τις μεταφορές εσωτερικές υδάτινους οδούς και ελπίζουμε ότι στις 17 Δεκεμβρίου θα ε, αποφασίσει το Συμβούλιο κάτι αντίστοιχο σε ό,τι αφορά για τους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν. Ας έρθω τώρα στα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών συγκοινωνιών. Νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα εξετάσουμε μέσα στα πλαίσια του μεγάλου αριθμού των επιβατών οι οποίοι πετούν κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το αριθμό των αεροπορικών εταιρεών. Αυξάνει συνεχώς μεν ο αριθμός των παραπώνων. Εμείς έχουμε λάβει ήδη 553 τέτοιες ε, ε, διατυπώσεις παραπώνων μόνο το Σεπτέμβριο σε σχέση με τον κανονισμό του 2004 αλλά η εφαρμογή του κανονισμού αυτού για τα δικαιώματα των επιβατών είναι καταρχήν ευθύνη των εθνικών υπηρεσιών έχουν καθοριστεί οι αρμόδιοι φορεί σε εθνικό επίπεδο, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού. Κάθε χρόνο αυτοί οι φορεί ε, λαμβάνουν περίπου 50.000 παράπονα, τουλάχιστον αυτό ήταν ο αριθμό για το 2008, κυρίως για τον κανονισμό του 261 του 2004. Το γεγονός ότι επαφίεται στην εθνική ευθύνη η εφαρμογή αυτού του κανονισμού δεν σημαίνει ότι η Κομισιόν δεν είναι πάρα πολύ ενεργή. Καταρχήν, η Κομισιόν οργανώνει τακτικά επαφές με εθνικούς φορείς εφαρμογής αυτού του κανονισμού, ώστε όχι μόνο να εφαρμόσετε ορθά αυτός ο κανονισμός, αλλά και με ένα ομοιόμορφο τρόπο σε όλο το μήκος, το πλάτος και το βάθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πολυμερείς επαφές, αλλά και διμερείς επαφές με μεμονωμένες εθνικές αρχές, και επίσης έχουμε οργανώσει δύο συνδιασκέψεις σε σχέση με τον κανονισμό 261 και σχεδιάσουμε να οργανώσουμε άλλη μια τέτοια συνδιάσκεψη στην αρχή του 2010. Ενδιαμέσως. Θα λάβει χώρα και μια ειδική συνάντηση σε δύο εβδομάδες στις 23 Νοεμβρίου με τους εθνικούς φορείς εφαρμογής που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή του κανονισμού 117 του 2006 για τα δικαιώματα των επιβατών με περιορισμένη κινητικότητα. Μια άλλη δραστηριότητα είναι η εκκίνηση μιας έρευνας τον προηγούμενο Μάρτιο από τον ε, Αντιπρόεδρο Ταγιάννη για να μπορέσουμε να εξετάσουμε καλύτερα τα στοιχεία σε σχέση με όλα τα προβλήματα τα οποία συνάπτονται με τις αποσκευές εναερίες μεταφορές τα τελευταία χρόνια η ανάλυση των απαντήσεων που λάβαμε έχει επιβεβαιώσει την ε, εντύπωση ότι σε απόλυτο αριθμό, σε ό,τι αφορά του απόλυτου αριθμού, υπάρχουν πραγματικά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Βάσει των στοιχείων που είναι διαθέσιμα, ο αριθμό των αποσκευών που καθυστερούν στα αεροδρόμια είναι περίπου 4,6 εκατομμύρια μεταξύ του Ιανουαρίου του 2008 και του Οκτωβρίου του 2008, δηλαδή σε μία περίοδο 10 μηνών. Έχουμε επίσης τρεις συνεχιζόμενες μελέτες, μία για την εφαρμογή του κανονισμού 261 και από και άλλες μελέτες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για μας, για να μας πληροφορήσουν σε σχέση με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, τη στιγμή που δεν υπάρχει υποχρέωση από την πλευρά των κατών μερών να μας δίνουν τακτικές ε, αναφορές. Η τρίτη μελέτη αφορά τα εθνικά συστήματα κυρώσεων, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη, για την εφαρμογή του κανονισμού 1107 για τα δικαιώματα των επιβατών. Και μετά από μια πρόσφατη έρευνα, θα ξεκινήσουμε και μια νέα μελέτη σε σχέση με το θέμα των αποσκευών. και θα ξεκινήσουμε μετά μια αχανή δημόσια διαβούλευση σε σχέση με τα δικαιώματα των επιβατών και η οποία θα περιλαμβάνει προφανώς και όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη μεταφορά των αποσκευών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι λοιπόν θα πρέπει από όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών χωρών να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία και θα είναι ιδιαίτερα καλόδεκτη και σημαντική η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή την έρευνα. Στις αρχές του 2010 η Κομισιόν θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης και θα οργανώσει και την διάσκεψη την οποία ανέφερα προηγουμένως για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Τέλος, όλες αυτές οι πηγές πληροφοριών, τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και τα πορίσματα των μελετών που συνεχίζονται θα είναι η βάση επί της οποίας η Κομισιόν θα εκδώσει μια ανακοίνωση το 2010 που θα καλύπτει όχι μονάχα την αξιολόγηση της ποιότητας εφαρμογής του τωρινού κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, αλλά θα είναι και η βάση για αξιολόγηση περαιτέρων μελλοντικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε ρυθμιστικό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. For the PPE. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντιβέρα από πλευρά ΣΕΛΚ. Ευχαριστώ που δεχθήκατε να μας παρουσιάσετε τα δικαιώματα των επιβατών στην Επιτροπή μα, Κυρία εκπρόσωπε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολλοί από όπως και πολλοί από του βουλευτές, έχω λάβει διαμαρτυρίε ε, πολιτών που του αρνήθηκαν την επιβίβαση παρόλο που αντιμετώπισαν σημαντικέ καθυστερήσει, δεν έλαβαν καμιά βοήθεια και δεν μπόρεσαν να αποφεληθούν από τα όσα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τι αποζημιώσει Και μετά το ισχύ αυτού του κανονισμού 261 του 2004 που καθορίζει σειρά δικαιωμάτων για τους επιβάτες αερογραμμών η προστασία των επιβατών εν γέννη βελτιώθηκε, όμως τα δικαιώματά τους δεν έγιναν σεβαστά πάντοτε και ο κανονισμός πολύ συχνά δεν εφαρμόζεται καλά. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα προέρχεται από τον ίδιο τον κανονισμό, αλλά εν μέρη προέρχεται από κάποιες χώρες και κάποιες ε, εφαρμοστικές αρχές, αρμόδιες αρχές που δεν επέβαλαν ε, τον νόμο. Και δεν είναι η μόνη υπεύθυνη αυτή η αλλά υπάρχει και ένα έλλειμμα από πλευρά του προσωπικού των εταιριών που είναι σε άμεση σχέση στο αεροδρόμιο με του επιβάτε και που δεν γνωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το προσωπικό, του ευρωπαϊκού κανόνε όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών εταιριών και δεν ε, πληροφορούν σωστά του επιβάτε γιατί βήματα μπορούν να κάνουν. Και αυτό μα το είπαν πάρα πολλοί ταξιδιώτε. Κυρία Χότσμαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προτίθεται να κάνει για να βελτιώσει την ενημέρωση των επιβατών και το πώ αντιμετωπίζει το αεροδρόμιο. Και έχω άλλο σχόλιο. Φαίνεται ότι ο κανονισμό του 2004 δεν καλύπτει όλε τι περιπτώσει Να δώσω ένα παράδειγμα, δύο παραδείγματα να δώσω. Το πρώτο, ένα επιβάτη που βλέπει να αναπρογραμματίζεται η πτήση του και αυτό δεν φαίνεται να καλύπτει το κείμενο και μετά έχουμε τον ταξιδιώτη που έχει μια ανταπόκριση με διαφορετικέ εταιρείε. Αν η καθυστέρηση τη πρώτη εταιρεία τον κάνει να χάσει την ε, άλλη πτήση, δεν τον αναλαμβάνει η εταιρεία αυτή που έχει καθυστερήσει γιατί τον υποχρεώνει ο κανονισμό, δεν του δίνει στέγαση και η δεύτερη δεν είναι υπεύθυνη διότι έφυγε στην ώρα τη η δεύτερη εταιρεία ανταπόκριση και καθυστέρησε ο επιβάτη. Οπότε υπάρχει ένα νομικό κενό που είναι επιζήμιο για τον πολίτη. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντιβέρακ. Ο κύριο Αλκαντράουι έχει το λόγο. Ομάδα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε, ευχαριστούμε κύριε Χάτμαν για αυτή την ε, παρουσίαση του θέματος, τη σύντομη παρουσίαση που κάνατε, που έχει σχέση με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών ε, εταιριών. Αναφερθήκατε στον ε, μεγάλο αριθμό των ενστάσεων που κατατίθενται, περίπου 50.000 το χρόνο, οι οποίες κατατίθενται στις εθνικές αρχές ε, πρόκειται για ένα αρκετά μεγάλο αριθμό και επισημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε διάφορα επίπεδα. Δηλαδή, αφενός έχουμε τις ε, καταγγελίες αυτές, ε, ενστάσεις καταγγελίες, ε, όπου υπάρχει ένας συνολικός αριθμός. Εσείς όμως ως Κομισιόν νομίζω ότι δεν έχετε σαφή εικόνα για το τι είδου καταγγελίες κατατίθενται. Φαντάζομαι μπορεί να διαφωνήσετε μαζί μου, αλλά εγώ πιστεύω ότι επειδή οι καταγγελίες αυτές ε, κατατίθενται συλλογικά στις εθνικές αρχές δεν έχουμε σαφή εικόνα του όλου θέματος. Ίσως ε, λοιπόν ε, θα ήταν καλύτερα οι καταγγελίες να λαμβάνουν συλλογική μορφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποκτάμε καλύτερη εικόνα. Και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον υπάρχει η τάση να κατατίθενται περισσότερες καταγγελίες σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Αν δηλαδή υπάρχει ένα γεωγραφικό χαρακτηριστικό όσον αφορά τις ε, καταγγελίες. Και κάτι άλλο επιτρέψτε μου να πω. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι υπήρξαν ε, περιπτώσεις ε, λογοκρισίας, ότι υπάρχει, υπάρχουν δυνατότητες κατάχρησης να γίνει δηλαδή κατάχρηση κυρίως ε, της ε, περίπτωσης ε, ανωτέρας βίας. Και ρωτώ λοιπόν, διερωτώ με και εγώ και ρωτώ και εσάς, μήπως θα είχε νόημα να κλείσουμε αυτά τα κενά, να μην αφήνουμε περιθώριο για λογοκρισία και να διατυπώσουμε τη σχετική νομοθεσία με πιο αυστηρό ύφο. Και τελευταία μου παρατήρηση κάποια στιγμή πρόκειται να έχουμε μία σαφή εικόνα σχετικά με την ε, εφαρμογή των κανονισμών που υπάρχουν ε, σε αυτόν τον τομέα για τα δικαιώματα των επιβατών ε, αεροπορικών εταιριών. Γιατί αν είχαμε μία σαφή εικόνα θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε τι ακόμα εκρεμεί τι πρέπει να ρυθμιστεί. Εσείς παραδείγματος χάρη δείξατε το θέμα των αποσκευών. Κάτι γίνεται από αυτού, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα που θα έπρεπε να ρυθμιστούν, ε, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η πλημμυρίδα των καταγγελιών και θα μπορούσε να μας βοηθήσει να γνωρίζουμε καλύτερα πού πρέπει να ξεκινήσουμε. Σε ευχαριστώ κύριε Καντράι, Πλανσάρ, για την άντε, κύριε Πλανσάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω ε, να προσθέσω τίποτα, ουδέν κενών υπό τον ήλιο. Και εγώ εδώ και εβδομάδες γνωρίζω ότι υπάρχει μια ολόκληρη πλημμυρίδα ε, καταγγελιών εις βάρος αεροπορικών εταιριών που ε, καταπατούν τα δικαιώματα των επιβατών. Δεν είναι ότι ο επιβάτης έχει πάντα δίκιο, αλλά κατά κανόνα έχει δίκιο. Εκείνο λοιπόν που ενδιαφέρει είναι να καλύψουμε κενά ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία. Ίσως ε, θα πρέπει να δούμε λιγάκι τι ερμηνεία μπορούμε να δώσουμε στα έγγραφα της ε, Κομισιόν, τα έγγραφα τα οποία η Κομισιόν επεξεργάστηκε από κοινού με τους ε, εμπλεκόμενους. Και εάν λοιπόν κατανοούμε καλά, τότε δεν είναι ότι το έγγραφο αυτό οδήγησε στο να μειωθεί ο αριθμός των καταγγελιών. Διερωτώμε λοιπόν τι θα γίνει στο μέλλον, γιατί το 2010 τελικά θα κατατεθούν θα εξαχθούν τα συμπεράσματα από άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί. Βεβαίως αυτή η διαδικασία μπορεί να ε, συνεχιστεί στο διηνεκές. Σε τελική ανάλυση όμως η Κομισιόν δεν μας λέει τίποτα το καινούριο, κυρίως εκεί όπου πρόκειται για την ομοθεσία. Υπάρχουν αυτά κενά, υπάρχει και ένα είδος ε, λογοκρισίας. Και εγώ διερωτώ με, θα πρέπει να περιμένουμε όλες αυτές τις ε, έρευνες, γιατί δεν είναι δυνατόν να μας αναφέρουν συνεχώς αυτό το γεγονός ότι γίνονται έρευνες. Στην Ιμπέρια, παραδείγματος χάρη, εκεί δεν πρόκειται για ένα επιβάτη, πρόκειται για εκατοντάδες επιβατών οι οποίοι τους λένε, στους οποίους λένε συνεχώς ναι, αλλά τελικά τίποτα δεν γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πάρει ποτέ αποζημίωση και με κατά πόσο η Κομισιόν μπορεί να παρέμβει στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ε, κυρία για Um, um, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έκθεσή σας, ε, η οποία πράγματι έπρεπε να έχει κατατεθεί εδώ και πολύ καιρό και είναι απολύτως απαραίτητη. Εγώ διαπιστώνω ότι τελικά τα δικαιώματα των επιβατών δεν βελτιώνονται όπως θα έπρεπε. Εγώ συγκεντρώνω στατιστικά δεδομένα για μένα, για τον εαυτό μου και κατά την τελευταία θητεία 17 φορές καθυστέρησε η ε, βαλίτσα μου και άλλοι αναφέρουν ακόμα και καθυστέρηση τριών μηνών. Αυτή έτσι είναι απλά μία δειγματοληψία που έκανα και επειδή περίμενα κι εγώ να δω τι θα γίνει με τη βαλίτσα μου, άκουσα ότι πάρα πολλοί άνθρωποι διαμαρτύρονται για το ότι ε, έχουν καταθέσει τέτοιου είδου περιπτώσει καταγγελίε για να ικανοποιηθούν ε, στα δικαιώματά του. Όμω η όλη η γραφειοκρατική διαδικασία είναι τεράστια, αποτρεπτική και γι' αυτό συνήθω παρετούνται. Αυτό ισχύει και για τα μαξίδια ε, για τα άτομα με αναπηρία πάρα πολλοί ανάπηροι μου έχουν στείλει διαμαρτυρίες για το θέμα αυτό και οποτεδήποτε εγώ τους έχω πει ότι θέλετε να, το, να παρακολουθήσουμε την υπόθεση μου λένε όχι δεν θέλουμε γιατί αν το κάνουν τότε πια η αεροπορική εταιρεία θα αρνηθεί να τους επιβιβάσει. Αλλά καταλαβαίνετε από ό,τι φαίνεται υπάρχει σε αεροπορικές εταιρείε ένας μαύρος κατάλογος των ανεπιθύμητων επιβατών οι οποίοι επιμένουν στην ε, ικανοποίηση των ε, δικαιωμάτων τους. Ίσως θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε λιγάκι αυτό γιατί εγώ ενημερώθηκα από επιβάτης ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Τώρα, σε κάτι πιο επίσημο επίπεδο θα ήθελα να μάθω. Τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε ε, σχετικά με αυτή την περίπτωση του denied boarding, της άρνησης ε, επιβίβασης ή ε, το ότι εμφανίζονται τεχνικές δυσκολίες και λήψεις σε πολύ λίγους επιβάτες αναφέρομαι στο κατά πόσον μπορούμε να θεωρήσουμε από τον αριθμό των καταγγελιών που κατατίθενται ότι ο αριθμός αυτός αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Γιατί σας είπα ότι υπάρχει η γραφειοκρατική διαδικασία που δεν επιτρέπει να είμαστε σαφείς στα συμπεράσματά μας. Παρακαλώ να το συμπεριλάβετε αυτό στη μελέτη σας. Πάρα πολλοί επιβάτες λένε δεν έχει κανένα νόημα να ξεκινήσω την όλη διαδικασία γιατί είναι τόσο χρονοβόρα, τόσο φθοροποιώσει η διαδικασία που στη τελική ανάλυση περισσότερη εργασία και κόπο μου κοστίζει από την αποζημίωση που θα πάρω. Τα κράτη-μέλη όσον αφορά την ε, μη ικανοποιητική εφαρμογή. Η διαδικασία της διαιτησίας, πώς μπορεί αυτή να λάβει χώρα. Αν δεν υπάρχει ανεξαρτησία, τότε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την αμεροληψία της διαιτησίας και πώς θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε την εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών όταν βλέπουμε ότι ε, σε κάποιες αεροπορικές εταιρείε, σε κάποια κρατημέλη δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Εγώ λοιπόν βλέπω να υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα όσον αφορά την ε, εφαρμογή και την ε, περίφημη enforcement, την επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών. Κάποια στιγμή όλα αυτά γίνονται νεκρό γράμμα. Γιατί τι γίνεται, κατατίθενται διαδικασίες, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει τίποτα από αυτόν. Και κάτι τελευταίο. Ένα σημαντικό σημείο στο θέμα των δικαιωμάτων των επιβατών είναι και να είναι σωστή και ε, ακριβής η αναφορά του ε, κόστους του ε, αεροπορικού εισιτηρίου. Είδατε τι γίνεται, μερικές φορές βλέπει κανείς το εισιτήριο για το Λονδίνο κοστίζει 99 ευρώ και τελικά όμως όταν πρόκειται να πληρώσει, καλείται κανείς να πληρώσει 130 ευρώ. Θα ήθελα λοιπόν να σκεφτούμε τι είδους μηχανισμός μπορεί να βοηθήσει για να μην παραμείνουν όλα αυτά νεκρογράμμα. Σας είπα ότι κάτι τέτοιο θα, θα οδηγήσει και ε, στο να αντιμετωπίσουμε εμείς πολλά προβλήματα. Τον τελευταίο καιρό διαπίστωσα ότι οι αεροπορικές εταιρείες ε, αντιμετωπίζουν ε, τον επιβάτη ως ένα αρνητικό, δυσάρεστο στοιχείο το οποίο καλούνται να μεταφέρουν και αυτό είναι μια κατάσταση απαράδεκτη. Κύριε Φώστερ, ευχαριστώ. <clears throat> Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επανήλθε σε αυτή την Επιτροπή όμως, επανήλθε για μια ενημέρωση για τον κανονισμό του 2004. Ήμουνα τότε μέλος και το θυμάμαι καλά τον κανονισμό. Πολύ λίγα στατιστικά μας δόθηκαν. Μιλήσαμε για 738 εκατομμύρια επιβάτες μετά αναφέρονται 553 έρευνε. Τι είναι μια έρευνα και τι είναι καταγγελία και τι είναι διαμαρτυρία. Μετά αναφερθήκανε 50.000 καταγγελίε και έρευνε. Αναγνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετώπισε προβλήματα για τη συλλογή πληροφοριών. Και πριν από αρκετά χρόνια είχαν πάρουν προβλήματα να πάρουν πληροφορίε από τα κράτη-μέλη, γιατί κάποια κράτη-μέλη συλλέγουν τι πληροφορίε του με πολύ καλύτερο τρόπο. Αλλά δεν έχει νόημα να επανέρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επιτροπή και να μα πετάει αυτά τα στοιχεία διότι αυτό που θέλουμε να ξέρουμε σαν μέλη της Επιτροπής είναι περί τίνος πρόκειται, τι συζητάμε. Ήταν πάρα πολύ καλός ο κανονισμός που θεσπίστηκε το 2004 και είναι λίγο φαϊνότερο ποιε είναι οι απαιτήσει των εταιριών και όλων των άλλων και τι επιτρέπεται να αποκτήσουν οι επιβάτες. Με εξαίρεση αυτών. Τι ξέρουμε. Ότι κάποιες αεροπορικές εταιρείε και πριν την νομοθεσία ήταν πολύ καλή μεταφορής και οι επιβάτες ήταν πολύ ευχαριστημένοι. Και τότε ο λόγος για τη θέσπιση του κανονισμού ήταν ότι υπήρχαν άλλες εταιρείε που δεν συμμορφωνόταν και δεν πρόσεχαν τους πελάτες τους. Γι' αυτό λοιπόν ε, φτιάξαμε αυτόν τον κανονισμό. Θεωρώ λοιπόν ότι παρόλες τις ελάχιστες πληροφορίες που μας δόθηκαν από εσά, κυρία μου, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρόλα αυτά έχουμε έναν κανονισμό. Δεν ερμηνεύεται σωστά δεν εφαρμόζεται σωστά. Πολλές εταιρείε κινούνται σωστά, αλλά κάποιες εταιρείε όχι. Πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι εταιρείε και να αντιμετωπίζετε αυτές οι εταιρείε που δεν συμμορφώνονται και που αντιμετωπίζουν άσχημα τους επιβάτες τους. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Είναι κατά πόσο ε, πρέπει να είναι ανάλογα τα μέτρα που θα λάβετε δεν είναι ότι δεν χρειάζεται να εξετάζουμε το θέμα που καιρού εις καιρών βεβαίως πρέπει να γίνεται, αλλά πιο επικοδομητικά, πολύ πιο επικοδομητικά. Και θα ήθελα να πω, Πρόεδρε, ότι η κυρία Λιχτανμπέργκερ σωστά έθεσε το θέμα της τιμολόγησης. Ξέρουμε ότι πολλοί μεταφορές έχουν πολύ καλές ιστοσελίδες. Όταν πάει κανείς σε ιστοσελίδα, ξέρεις ακριβώς ποιο είναι το συνολικό ποσό πριν, πληρώσει πριν φτάσει στη σελίδα. Αλλά Λοιπόν, πρέπει να περάσει άριστο σελίδε, τουλάχιστον 20-23 σελίδε μέχρι να βρει το τελικό ποσό πρέπει να καταβάλει. Κάποιε εταιρείε δίνουν σωστέ πληροφορίε, κάποιε όχι. Οπότε υπάρχει ανισότητα εδώ και χρειάζεται πολλέ διευκρινήσει. Προτείνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιστρέψει ξανά στην Επιτροπή αργότερα με λεπτομερέστατες πληροφορίες περί της καταστάσεως. Και μετά μπορούμε να δούμε κατά πόσο χρειάζεται άλλη ανακοίνωση, άλλος κανονισμός, μια προσθήκη, κάτι άλλο κάποτε στο μέλλον. Λοιπόν, από την δική μας ομάδα αυτό είναι που έχουμε να προτείνουμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Κόλσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι υπάρχουν 50 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν δικαιώματα τα οποία βάσει του κανονισμού τουλάχιστον είναι εγγυημένα. Στα χαρτιά. Από ό,τι έχουμε δει όμως υπάρχει ένας αριθμός προβλημάτων. Τα άτομα τα οποία έχουν αναπηρίες αντιμετωπίζουν αρνητικές διακρίσεις εναντίον τους. Υπάρχει έλλειψη ίσης μεταχείρισης όταν τα άτομα αυτά με αναπηρίες ταξιδεύουν. Το πρώτο μου ερώτημα είναι ποια είναι η πρόθεση της Κομισιόν για να σταματήσει αυτή η διάκριση των ατόμων που έχουν αναπηρίες, ώστε να υπάρχει πράγματι σεβασμός των δικαιωμάτων τους και σεβασμός της ισότητας μεταχείρισής τους εναντί των άλλων επιβατών. Για μένα το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο την χάνει η ερμηνεία σε αυτός ο κανονισμός. Δίδονται διαφορετικές ερμηνείες. Ένας από, μια βουλευτής ήδη αναφέρθηκε στο θέμα των ε, ε, αναπηρικών πολυθρονών, των αμαξιδίων. Αυτό δεν είναι αποσκευή. Αλλά πολλές αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν τα αναπηρικά καροτσάκια αυτά σαν να είναι κομμάτια, σαν να τμήματα των αποσκευών ενός ατόμου. Πολλές φορές κάποιος ο οποίος χρειάζεται την αναπηρική πολυθρόνα αναγκάζεται να τη στερηθεί για μια ολόκληρη μέρα. Λέει επίσης ο κανονισμός ότι μπορεί κανείς για ορισμένους λόγους να αρνηθεί την πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία σε ορισμένες ε, πτήσεις. Η, μια ισπανική ε, εταιρεία χρησιμοποίησε αυτό σαν ε, πρόσχημα για να αρνηθεί την επιβίβαση σε έξι επιβάτες οι οποίοι ήταν κοφοί. Θα ήθελα λοιπόν να καταλάβω ποια είναι η σωστή ερμηνεία στα θέματα αυτά και πώς η Κομισιόν προτίθεται να δράσει και να εξασφαλίσει ότι ασκείται πάντα η σωστή Υπάρχει πάντα η σωστή ερμηνεία αυτού του κανονισμού σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, νομίζω ότι προτού εγκριθεί ένας άλλος κανονισμός, θα πρέπει να ακουστεί και η άποψη των εκπροσώπων των ατόμων με αναπηρίες. Ευχαριστώ. <coughs> Ευχαριστώ πολύ κύριε Κόλσα. Ε, ο Αντιπρόεδρος έχει το λόγο. Κύριε Ζήκε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν η οποία μας παρουσίασε το θέμα αυτό του κανονισμού. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες βέβαια. Αυτό φαίνεται και από τον αριθμό των παραπώνων και των καταγγελιών που είναι σημαντικός. Το ερώτημα τώρα είναι αν μπορούμε να έχουμε κάποια εικόνα για τον αριθμό των καταγγελιών οι οποίες ευδοκιμούν κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή που δίδουν, συνέ, δίδουν λαβή σε θετικές συνέχειες από την πλευρά των αρμοδίων αρχών. Δεύτερον, γνωρίζουμε πόσες από αυτές τις καταγγελίες καταλήγουν στα δικαστήρια, σε ένδικες διαδικασίες και ποια είναι η συνέχεια που δίνεται στην περίπτωση αυτή. Και το τρίτο ερώτημα είναι ποια μέσα κατασταλτικά, ποια μέσα, εν επιβολής έχει η Κομισιόν στη διάθεσή της για να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός. Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κανονισμοί οι οποίοι είναι όλο και πιο λεπτομερείς, αλλά υπάρχουν όλο και περισσότερες καταγγελίες. Φαίνεται λοιπόν ότι οι κανονισμοί τελικά δεν υποχρεώνουν τις εταιρείε να εφαρμόσουν το περιεχόμενο του κανονισμού. Επομένως είναι σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι η συνέχεια που δίνεται στις καταγγελίες, πόσες από αυτές καταλήγουν στα δικαστήρια, ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των διαδικασιών και πρέπει να σταματήσουμε να εργαζόμαστε μόνο σε ένα θεωρητικό επίπεδο και να δούμε στην πράξη τι σημαίνουν όλα αυτά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θα ήθελα να αφαιρθώ σε αυτά που είπε η κυρία Ρικέ. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτά τα οποία μπορούμε να ρυθμίσουμε εδώ για τους επιβάτες μέσω κανονισμού, πράγματι να το πράξουμε, να προωθήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία γιατί ε, κάτι τέτοιο το περιμένουν και οι πολίτες. Υπάρχουν ε, πάρα πολλοί κανονισμοί, όμως ε, πρέπει να πούμε ότι ως επιβάτης, αναφέρομαι σε εκείνον που δεν πετάει κάθε μέρα, ο κανονικός, ο απλός επιβάτης δεν είναι σε θέση να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνουν γνωστά τα δικαιώματα και κατά δεύτερον να έχουμε κατά νου ότι θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ε, στους ε, ε, πολίτες τι ακριβώς πρέπει να κάνουν για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Ξέρω παραδείγματος χάρη μια περίπτωση όπου τα δικαιώματα μπορεί κανείς να τα διεκδικήσει μέσα από οργανισμούς προστασίας καταναλωτών. Γνωρίζει ότι είναι πολύ δύσκολο να καταφύγει κανείς κατά μιας αεροπορικής γιατί κάτι τέτοιο να έχει και το στοιχείο του κινδύνου ως προς το κόστος. Θα ήταν λοιπόν σωστό για τους επιβάτες αν μπορούσαμε να τους δώσουμε ένα όπλο, ένα εργαλείο για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Προφανώς και αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά παρόλα αυτά εγώ θεωρώ ότι πρέπει και εμείς να σκεφτούμε πάνω στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει άλλος ε, στον κατάλογο του Προέδρου. Να πω ότι στην κυρία Χούτμαν σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας. Να πω εξ αρχής κάτι. Κάτι που δεν θέλω να δω. Δεν θέλω το Κοινοβούλιο να επιμένει επί κανονισμών που κάνουν λιγότερο ασφαλή τις πτήσεις από ό,τι είναι τώρα. Ξέρουμε βέβαια ότι οι πτήσεις είναι πολύ ασφαλείς μεταφορές. Δεν θέλω οι πιλότοι να βρεθούν σε δύσκολη θέση, να πρέπει να αποφασίσουν κατά πόσο πρέπει να πετάξουν ή να πληρώσουν αποζημίωση. Πρέπει να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία. Ό,τι και να κάνουμε που θα απορρέει από τον κανονισμό 261. Η εντύπωση που σχηματίζω κάθε φορά είναι ότι υπάρχει σαφώς έλλειψη ενημέρωσης των επιβατών. Δεν ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά τους όταν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα καθυστέρηση, ακύρωση και σίγουρα υπάρχει σαφή έλλειψη γνώσεων από πλευρά προσωπικού αεροπορικών εταιριών και κυρίω προσωπικού εδάφου όταν προκύπτει ένα πρόβλημα σχετικά με τις δικές τους υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις που απορρέουν τον κανονισμό. Τώρα, εάν αυτό είναι δικό μας πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, διότι δεν επιμένουμε στην κατάλληλη κατάρτισή τους ή αν είναι πρόβλημα των αεροπορικών εταιριών, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν με ενδιαφέρει ποιο θέλει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βρεθεί λύση, ούτω ώστε το προσωπικό εδάφους να ξέρει ποιες είναι οι υποχρεώσεις του βάσει του κανονισμού. Ξέρω τα θαύματα χρειάζονται κάποιο χρόνο, διότι το προσωπικό εδάφους πολύ συχνά δεν ξέρει ότι έχει καθυστερήσει καν οι πτήσεις. Συνήθω οι επιβάτες τους λένε ότι καθυστερεί και ούτε ξέρουν που πήγε η πτήση κλπ. Και εγώ στο Μάντσεστερ την περασμένη εβδομάδα αυτά πέρασα. Τόσο πολλά. Κάτι άλλο πρέπει να εξετάσουμε. Οι καθυστερήσεις είναι ο άλλος τομέας. Η κυρία Χάνες Πλασέ είπε ότι πρέπει να δούμε ποιες καταγγελίες, ποια είδη καταγγελιών είναι οι περισσότερες ακυρώσεις ή καθυστερήσεις. Εγώ υποψιάζομαι περισσότερο πρόβλημα με καθυστερήσεις θα έχουμε, διότι μαζί με τις καθυστερήσεις έχουμε και άλλο θέμα το, κα, καφέ, το γεύμα κλπ. πρέπει να προσφερθεί και θα είναι χρήσιμο να υπάρχει τομεακή κατανομή των στοιχείων. Όχι μόνο ότι πρόκειται περί καθυστερήσεων, ακυρώσεων κλπ. Αλλά επίσης ποιες αεροπορικές εταιρείες δημιουργούν τα περισσότερα προβλήματα. Είναι τα charter, ε, είναι οι κανονικές, τα κανονικά δρομολόγια, τακτικές, τα, τακτικά δρομολόγια ή εταιρείε οι ε, ή περιφερειακές. Αν έχουμε τις πληροφορίες αυτές μπορούμε να προχωρήσουμε. Μπορούμε να εξετάσουμε καλύτερα τα αίτια. Επιτρέψτε μου να πω ότι επίσης και το θέμα είναι της αλλαγής του δρομολογίου. Αλλάζουν μόνο Μπορεί να κάθεσαι πέντε ώρες στο αεροδρόμιο εσύ, να περιμένεις για την επόμενη πτήση τους και προτιμάς να κάνεις αυτό παρά να πάει στο αεροπλάνο που πάει Βρυξέλλες το οποίο θα σε πήγαινε σε άλλη πτήση που θα φύγει μόλις σε μία ώρα για κάπου αλλού. Δηλαδή να σε, να σε πάνε μέσω άλλου δρομολογίου στον προορισμό σου. Α, αλλαγή διαδρομή δεν είναι ότι σε πάει με τη δική σου αεροπορική εταιρεία και σε φτάνει στον προορισμό σου μέχρι άλλη, μέσω άλλη διαδρομή, αλλά σε πάνε με άλλη αεροπορική εταιρεία και δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Να πω τρία πράγματα. Η τιμολόγηση αναφέρθηκε. Και έχουμε προβλήματα. Πετάξτε στο Δουβλίνο για ένα ευρώ σου λένε. Εγώ δεν πιστεύω ότι πέταξε κανείς του και πήγε στο Δουβλίνο με ένα ευρώ. Και αυτό πρέπει να το δούμε και μετά η ασφάλιση. Και οι ομάδες των ηλικιωμένων δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλικιωμένοι όσον αφορά την ασφάλιση που μπορούν να πληρώσουν για τα ταξίδια τους. Είτε για διακοπές πηγαίνουν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Γιατί το αναφέρω αυτό. 20 χρόνια είμαι στο Κοινοβούλιο. Και στο περισσότερο διάστημα εγώ επέμενα ότι χρειάζεται ένα νέο πακέτο για τα, για τα ταξίδια, νέα οδηγία που θα συνδέεται με αυτά που κάνουμε για τον κανονισμό 261. Αλλά ποτέ δεν δημιουργήθηκε αυτή. Έχουμε τα προβλήματα με τις ασφαλίσεις. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να πληρώσουν τα ασφάλιστρα για να ταξιδέψουν. Ο κύριος Κόζα αναφέρθηκε στα άτομα με αναπηρίες και άλλοι αναφέρθηκαν σε αυτό. 2009 είμαστε τώρα και έχουμε μπει σχεδόν στο 2010. Δεν είναι απέσιο, φρικτό που δεν μπορούν να πετάξουν κάποιοι άνθρωποι, τους αρνούνται το δικαίωμα να πετάξουν ή δεν μπορούν να ταξιδέψουν με οποιοδήποτε μέσο λόγω αναπηρίας. Αυτό είναι βικτοριανής εποχής. Δεν είναι κάτι το οποίο έπρεπε να συμβαίνει το 2010. Και ξέρω και υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που χρειάζεται οξυγόνο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει κανεί οξυγόνο Μπορεί να χρησιμοποιήσει το οξυγόνο του λένε στο αεροπλάνο, να χρησιμοποιήσει το δικό μας και θα πληρώσετε τόσα χύψη ωμέγα. Πρέπει να επανεξετάσουμε τον κανονισμό 261. Θα πρέπει να καλυφθούν τα κένα. Και το θέμα της ανώτερης βίας. Μας βοήθησε σχετικά το δικαστήριο όταν αποφάσισε ότι αν φύγει ένα φτερό από ένα αεροπλάνο αυτό δεν είναι ανώτερα βία εμείς το ξέραμε αυτό από την αρχή. Και δυστυχώς κάποιε από τις εταιρείε το ξέρανε. Και πρέπει να τονίσουμε αυτό που τόνισε η κυρία Φώστερ. Δεν κυνηγάμε τους καλούς. Αυτούς που έπρεπε να κυνηγάμε είναι οι κακοί. Και για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε στατιστικά στοιχεία, χρειαζόμαστε στοιχεία και γεγονότα, στοιχεία συγκεκριμένα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον αυτόν τον κανονισμό. Είναι δική σας ευθύνη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μας δώσετε αυτά τα στοιχεία και τις πληροφορίες. Ίσως έχετε κάποιες απόψεις για τις ιδέες που έχετε στο μυαλό σας. Μην αφήσετε σε εμά τα, τα θέματα νομοθεσίας. Μάλλον αφήσετε την νομοθεσία σε εμά. Εμείς μπορούμε να θεσπίσουμε νομοθεσία μόνο μας τα στοιχεία. Πού πρέπει να στοχεύσουμε. Σε επίπεδο 100 μελών πρέπει να στοχεύσουμε σε επίπεδο κάποιων αεροπορικών εταιριών. Ποιου πρέπει να βάλουμε στο στόχαστρο. Πρέπει να μα δώσετε τα πυρομαχικά. Και πιστέψτε με ότι αν μα δώσετε τα πυρομαχικά, εμεί τα πυροβολήσουμε. Καλώ. Κύριε Ρούτμαν, θέλετε να απαντήσετε, κόσμο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Yes, Mr. Βεβαίω, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα σχόλια τα οποία άκουσα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τονίσω ότι πράγματι υπάρχει ένα χάσμα πληροφορίας, μια έλλειψη πληροφορίας. Και γι' αυτό εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή την αχανή, την εκτενή πληροφοριακή εξαρτία που θα καλύψει τις αεροπορικές εταιρείες, τα αεροδρόμια και τους επιβάτες. Αυτό νομίζω θα βελτίωσει την κατάσταση. Όταν τώρα πρόκειται για τα τον ε, ε της αλλαγής ή των προβλημάτων των ανταποκρίσεων, τα προβλήματα των ανταποκρίσεων. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα καλυφθούν από τη δημόσια διαβούλευση που θα ξεκινήσουμε εμείς. Επομένως θα αποκτήσουμε πληροφορίες για τα θέματα αυτά, επί τη βάση των οποίων λοιπόν θα μπορέσουμε εμείς να σας πούμε κατά πόσο είναι απαραίτητο να υπάρξει μια τροποποίηση του κανονισμού για να καλυφθούν και αυτά τα νέα θέματα. Επίσης, όπως είπα προηγουμένως, το γεγονός ότι ο κανονισμός δεν περιλαμβάνει κάποια υποχρέωση εκθέσεων, παροχής εκθέσεων από τα κράτη-μέλη, αυτό οδηγεί σε προβλήματα για να μπορέσουμε να συλλέξουμε τα σωστά στοιχεία σε σχέση με την εφαρμογή του κανονισμού. Όπως ξέρετε, η αρχική πρόταση για τα λεωφορεία και τα πούλμαν είχαμε περιλάβει και μία υποχρέωση να υπάρχουν από τα κρατη και τους αρμόδιους φορείς εκθέσεις γιατί είχαμε πράγματι διδαχθεί αυτό το οποίο έπρεπε. Ο κ. Αλκαουντουρί έθεσε το ερώτημα της τυπολογίας των παγαπώνων. Μπορώ λοιπόν να σας πληροφορήσω ότι η κύρια πηγή συμβάντων που οδηγούν σε καταγγελίες, σε παράπονα, είναι η ακυρώσεις πτήσεων. Οι ακυρώσεις πτήσεων είναι περίπου 34,6% όλων των συμβάντων τα οποία ε, καταγράφονται μέσω παραπώνων. Η καθυστερήση των πτήσεων είναι πολύ κοντά με 32,5% των συμβάντων η άρνηση επιβίβασης 9,3% των συμβάντων και τα προβλήματα με τις αποσκευές είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. 5,4 απώλειες αποσκευών, 1,8% η βλάβη των αποσκευής, αποσκευές, 1,3% απώλεια αποσκευών. Υπάρχουν βέβαια και θέματα και τα οποία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, θα παίξει κάποιο ρόλο στην, ερμηνεία αυτού του κανονισμού. Είχαμε δύο αποφάσεις του δικαστηρίου που ερμήνευσαν καταρχήν την έννοια της πτήσης και δεύτερον την έννοια των εκτάκτων περιστάσεων της ανωτέρας βίας και το αναφέρω αυτό γιατί υπάρχουν πολλές φορές ε, για τεχνικούς λόγους καθυστερήσεις όπως αυτές που ανέφερε η κυρία Λίχτεμπεργκ διευκρίνησε εκεί το δικαστήριο ότι αυτές δεν αποτελούν έκτακτες περιστάσεις και επομένως εμπίπτουν στην φυσιολογική εφαρμογή του κανονισμού. Για το θέμα της επιβολής του κανονισμού. <clears throat> Πρέπει να επαναλάβω ότι υπάρχουν εθνικοί φορείς επιβολής και επομένως αυτή είναι αρμόδια για την επιβολή και την εποπτεία της εφαρμογής του κανονισμού. Στη συνέχεια, τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για την σωστή λειτουργία αυτών των φορέων παρακολούθησης σε εθνικό επίπεδο. Στο πρώτο επίπεδο λοιπόν των εθνικών φορέων εφαρμογής υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής <clears throat> επιβολής μάλλον κυρώσεων και μπορώ να σας πω ότι σχεδόν όλα τα κρατημέλη έχουν αναφέρει ότι επέβαλαν κυρώσεις σε κάποιες αεροπορικέ εταιρείες. Δεύτερον, αν δούμε ότι οι εθνικοί φορείς επιβολή δεν κάνουν σωστά τη δουλειά του, τότε η Κομισιόν μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία λόγω παραβάσεω εναντίον του αντίστοιχου κράτου μέλου. Αλλά αυτό θα πρέπει να βασιστεί σε μια κατάδειξη, σε μια διακρύβωση μιας κατασυρώη αποτυχίας αυτών των φορέων να κάνουν το, τη δουλειά του, να παίξουν το ρόλο του για το θέμα αυτό της διαφάνειας σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση των πτήσεων που έθιξε και η κυρία Λίχτεμπερ και η κυρία Πλάσνικ. Αυτό καλύπτεται από τον κανονισμό 108 του 2008, ο οποίος ετέθησε εφαρμογή <clears throat> πέρσι. Επομένως, πιστεύω ότι η κατάσταση αυτή θα βελτιωθεί με την εφαρμογή. Εφαρμογή αυτού του κανονισμού υπάρχουν βέβαια και ορισμένα ζητήματα τα οποία δεν καλύπτονται από τον καθορισμό αυτό, όπως παραγωγός χάρη τα πρόσθετα τέλη για τις αποσκευές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουμε στην δημόσια διαβούλευση, την οποία, όπως σας είπα, θα ξεκινήσουμε σύντομα. Τι άλλο, τι άλλο. Για τα αριθμητικά στοιχεία, βεβαίως, όπως ανέφερα, έχουμε πολλές μελέτες πέραν αυτών τις οποίες εγώ προανέφερα δύο μελέτες της ΕΑΖΑ, οι οποίες είναι σε εξέλιξη και θα επανέλθω, πιστεύω, με περισσότερα στοιχεία που μπορούμε να σας δώσουμε για όλες αυτές τις δραστηριότητες. Είναι σαφές ότι η εφαρμογή του κανονισμού δεν είναι τέλεια, αλλά έχουμε συνεργαστεί από πολύ κοντά με του βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή. Θα θυμάστε ότι εξεργήσαμε στην Επιτροπή σας ότι είχαμε μια πολύ στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τους βουλευτές για να έχουμε παραδείγματος χάρη κοινά ερωτηματολόγια για την υποβολή παραπώνων, τα οποία διευκολύνουν τη διαδικασία. Εξετάσαμε επίσης αν θα μπορούσαμε να έχουμε κοινά ερωτηματολόγια για τις ε, υπόλοιπες καταγγελίες και θα έπρεπε επίσης να σας αναφέρω ότι και από την πλευρά των επιβατών δεν είναι όλοι οι επιβάτες ικανοποιημένοι, αλλά και από τις αεροπορικές εταιρείες υπάρχουν πολλά παράπονα ότι ο κανονισμός αυτός είναι ιδιαίτερα αυστηρός με τις αεροπορικές εταιρείες. Ίσως η αλήθεια βρίσκεται και από τι δύο πλευρέ, Αλλά κύριε Πρόεδρε, η Κομισιόν κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο με του πόρου που έχει στη διάθεσή τη και θα είμαστε πάρα πολύ ενεργοί και στο μέλλον για να βελτιώσουμε την κατάσταση στο θέμα αυτό και όπω είπα και στην αρχική μου παρουσίαση, του χρόνου θα δημοσιεύσουμε μια ανακοίνωση η οποία θα βασίζεται σε όλε τι πληροφορίε οι οποίε θα συλλεγούν από τι διαβουλεύσει, τι συναντήσει με ευρωβουλευτέ και άλλου εμπλεκόμενου. και επομένω, αν είναι απαραίτητο, θα υπάρξει μια διαδικασία τροποποίησης του κανονισμού, ακόμα και πιθανώς πρόταση για νέα νομοθετήματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ λέει και ο, ο Πρόεδρος. Υποψιάζομαι ότι κάποιοι θα θέλανε να επανέλθουν στη συζήτηση. Θα είμαι πάρα πολύ λοιπόν αυστηρός. Αν θέλετε να επανέλθετε, θα πρέπει να είστε πάρα πολύ σύντομοι. Κυρία Πλάσνικ, Μπόσνικ και Λίχτεμπεργκ. Γιατί Νομίζω ότι πολλά ερωτήματα δεν απαντήθηκαν τελικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Γνωρίζω πολύ καλά ότι η Κομισιόν έχει δραστηριοποιηθεί στο θέμα αυτό και το εκτιμώ ιδιαίτερα, αλλά αυτό που με εκπλήσει είναι ότι υπάρχουν κάποιε περιπτώσει στα δικαστήρια, αλλά στη τελική ανάλυση δεν είναι ένδειξη αδυναμία εκ μέρου μα ότι αφήνουμε την νομοθεσία στα χέρια των δικαστήριων. Γιατί δεν θέλουμε εμεί να εξηγιάνουμε της, ε, την νομοθεσία και να μην αφήνουμε περιθώριο λιγμών για τους επιβάτες. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να στραφούμε στα δικαστηρία, θα πρέπει εμείς να επιληφθούμε τις νομοθεσίες, κάτι που είναι δική μας δουλειά. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω με, σε σχέση με αυτά που έγιναν κατά το παρελθόν. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει κανείς ε, να διεκδικήσει τα δικαιώματά του είναι να μην ε, υπάρξει κάποια νόθευση αυτών των δικαιωμάτων. Και γι' αυτό είπαμε και πολύ ότι υπάρχουν κενά. Η κυρία Φώστερ, πρόεδρε, θα ήταν χρήσιμο στο μέλλον όταν έρθει η Κομισιόν να ξαναστήσει για ένα τέτοιο θέμα ή οτιδήποτε άλλο να μας έχει δώσει ένα ενημερωτικό δελτίο για το τι πρόκειται να πει. Αυτό μας το δώσει πριν από τη συνάντηση με λεπτομέρειες για να μπορούμε να ενημερωθούμε. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι σε σχέση με τις ε, πληροφορίες που είπατε εσείς κύριε Πρόεδρε για την ε, αναδιαμόρφωση της ε, πτήσης και για περιπτώσεις όπου οι εταιρείε λένε ξέρετε δεν μπορείτε όμως να πάτε με την άλλη εταιρεία γιατί δεν είναι δική μας και δεν έχουμε συμφωνία μαζί τους. Κοιτάξτε, αν ασκήσει κανείς πίεση να ξέρετε ότι μπορεί ο επιβάτης να πάει σε άλλη εταιρεία. Μερικοί όμως δεν το λένε και αυτό λέει ο κανονισμός όταν εμείς τον εκπονήσαμε το 2003. Η κυρία Λιχτενμπέργκα. Έχω μία ερώτηση, δηλαδή συγκεκριμένα την εξή. Αρκεί να κάνουμε μόνο, να προβούμε μόνο σε ανακοίνωση όταν βλέπουμε ότι κατ' ουσίαν δεν έχουμε καμία δυνατότητα πρόσβαση σε δεδομένα ή ότι είμαστε αναγκασμένοι να θέσουμε σε εξωτερικούς μελέτες κάτι το οποίο θα έπρεπε να το κάνουν τα ίδια τα κράτη-μέλη και να στείλουν τις μελέτες αυτές στην Κομισιόν. Η ε, αερομεταφορίας θεωρείται ανέκαθεν ο τομέας εκείνος όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται τα μάλα. Αν τώρα όλα αυτά γίνονται στην πλάτη των επιβατών, καταλαβαίνετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της ε, δυσφημείται. Θα πρέπει λοιπόν να το έχουμε κατά νου αυτό και γι' αυτό ερωτώ ε, μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω και όχι να περιοριστούμε σε μια απλή ανακοίνωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω, με εκπλήσει λιγάκι το γεγονός ότι η Κομισιόν εξακολουθεί να διστάζει ε, να καταθέσει μια κοινή πρόταση. Αυτά όλα δεν είναι καινούρια. Ε, τέτοιου είδου ανάλυση είχε γίνει ήδη πριν από δύο χρόνια όταν κάναμε τότε την ανάλυση της νομοθεσίας και τότε είχαμε πει ότι καταρχήν θα προβούμε σε ανακοίνωση, μετά θα γίνουν οι αναλύσεις και τώρα ακούω πάλι τα ίδια και τα ίδια. Εγώ περιμένω από την Κομισιόν συγκεκριμένα μέτρα τα προβλήματα τα γνωρίζουμε, έχει γίνει συζήτηση, καλό είναι που γίνεται, αλλά τα κενά θα πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστούν. Και θα πρέπει να γίνει και κάτι όσον αφορά τους αριθμούς και την ερμηνεία των αριθμών. Γιατί εντάξει, καλά τους αναφέρετε τους αριθμούς, όμως πρόκειται κατ' ουσίαν μόνο για τις καταγγελίες που λαμβάνετε εσείς. Εγώ έτσι κατάλαβα. Όμως οι 50.000 καταγγελίες που κατατίθενται στα κράτη-μέλη, επ' αυτών δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν έχουμε ιδέα περί τίνος πρόκειται. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να επιληφθούμε εκ νέου του θέματος. Ο κύριος Wash. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν συντομία. Θεωρώ δεδομένο ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα των μελετών. Αλλά έχουμε νομίζω αρκετά στοιχεία για να μπορέσουμε να σκεφτούμε για προτάσεις τις οποίες ε, θα μπορούσε να υποβάλει η Κομισιόν. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να κάνουμε μελέτες, αλλά έχουμε αρκετά πρακτικά στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα λοιπόν να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των ε, επιβατών αεροπορικών γραμμών και φυσικά το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από την, ε, για να διατηρήσει τα δικαιώματα των ε, πολιτών. Θα ήταν λάθος λοιπόν να έχουμε λαθασμένα εκτελεστικά μέτρα οι μέτρα τα οποία τα καθυστερούμε στην εφαρμογή τους ή τα νερώνουμε κατά κάποιο τρόπο και δεν τους δίνουμε τη σωστή εφαρμογή. Κύριε Χούλετ, νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε ότι γενικά οι βουλευτές δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με τον τρέχοντα κανονισμό. Το λέω με διπλωματικό τρόπο όσο μπορώ και προσβλέπουν σε περισσότερη δράση από την πλευρά τη Κομισιόν. Αλλά για να είμαι και δίκαιος προς τον κύριο Κόζα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των ατόμων με αναπηρίες. Σας δίνω λοιπόν το λόγο και πάλι. Yes, thank you, Mr. President. Um, I mean, on the... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά το θέμα του προβλήματος ερμηνείας, το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ερμηνεύει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο σύνολό του και στις διαπραγματεύσεις για, τον κανονισμό, για τους κανονισμούς Ευρωπαϊκής Ενώσεως καμιά φορά έχουμε επικοδομητικές αμφισημίες όπως αποκαλούνται και οι συζητήσεις επί των ε, κειμένων ήταν πάρα πολύ δύσκολοι. Και δεν είναι σίγουρο ότι μια νέα συζήτηση προς διευκρίνηση των ενιών θα οδηγήσει σε καλύτερο κείμενο. Αν ο νομοθέτης δεν συμφωνεί, δεν θα υπάρχει περισσότερη σαφήνεια και το δικαστήριο κάνει έξοχη δουλειά διευκρινίζοντας τις έννοιες με τρόπο ο οποίος είναι πολύ ικανοποιητικό για το Κοινοβούλιο. Τώρα κατά πόσο αρκεί η ανακοίνωση είπα ότι η ανακοίνωση θα υποβάλει κάποιες νομοθετικές προτάσεις. Όπως ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε καλύτερο προγραμματισμό σαν αφορά κανονισμούς και υποχρεωνόμαστε να έχουμε σωστές πληροφορίες, πληροφορίες και στοιχεία για να γίνει σωστή αξιολόγηση αντικτύπου των προτάσεων και ήδη εξήγησα γιατί έχουμε πρόβλημα στοιχείων, που είναι αδυναμία αυτή βέβαια του κανονισμού. Ξέρουμε όμως ότι στις διαπραγματεύσεις για τα λεωφορεία και τα πούλμαν είχαμε πρόβλημα να πείσουμε τα κράτη-μέλη στις ομάδες εργασίας να υπάρχει σωστή ενημέρωση και υποβολή αναφορά στον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού. η Το θεωρούσαν μεγάλο διοικητικό άχθος. Εμείς επιμείναμε πολύ προφανώς να παραμείνει η διάταξη στο κείμενο αλλά ενδεχομένως ίσως αυτή είναι μια αλλαγή που θα πρέπει να επιφέρουμε στο κείμενο σχετικά με τις ε, αερομεταφορές. And for the second time, <laughs> Δεύτερη φορά. Άνθρωποι με αναπηρίες, σας παρακαλούμε. Are we really telling people with Λέμε θα προετοιμάσουμε μια ανακοινωσούλα για εσά άτομα με αναπηρία. αυτό του λέτε. Απάντηση. Όπως ήδη είπα, καλύπτεται αυτό από τι μελέτες που έχουν γίνει. Θα γίνει η συνάντηση επ' αυτού του θέματος στις 23 Νοεμβρίου με όλους τους φορείς των κρατών μελών και θα παρουσιάσουμε σχετικώς πρόταση του χρόνου και θα δούμε κατά πόσο υπάρχουν κάποια κενά στον κανονισμό και κατά πόσο χρειάζονται νέες διατάξεις σχετικά με τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Λυπούμε που ψάχνω τόσο πολύ του χρόνου πότε, Ιανουάριο του χρόνου, Δεκέμβριο του χρόνου. Διότι είναι επίγον πρόβλημα αυτό. Τώρα αυτό προσπαθούν να σας κάνουν να καταλάβετε τα μέλη. Αν μου πείτε Δεκέμβριο, 31 Δεκεμβρίου του 2010 θα στενοχωρηθώ λιγουλά και αν μου πείτε 1 Ιανουαρίου θα πω ότι είστε υπέροχοι. Μπορεί να δώσετε κάποια ένδειξη χρονική. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω ποιος θα είναι επίτροπος του χρόνου. Θα είναι νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη φάση να γνωρίζουμε πότε θα έχει προγραμματιστεί αυτή η ανακοίνωση. Σίγουρα θα είμαστε έτοιμοι το καλοκαίρι, μέχρι το καλοκαίρι. Δεν ξέρω όμως αν θα γίνει κάποιος αναπρογραμματισμός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Κόζα, προσπάθησα όσο μπορούσα. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Καλώς σας ευχαριστώ. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα όσο μας αφορά των συντονιστέ επιθυμία να συζητηθεί το θέμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από τις συστάσεις που υθετήσαμε στην έκθεση Σαβαρή στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου κατά πόσο είναι η κακή μέρα της κυρίας Χόπμαν δεν ξέρω αλλά είναι υπεύθυνη η κυρία Χόπμαν και για αυτό το θέμα Οπότε κυρία Χούτμαν έχετε το λόγο και για το σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα. Yes, thank you, Mr. President. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα την υποστήριξη που μας προσέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Εμείς, μισό λεπτό λέει ο Πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, αν έχει την καλοσύνη, αν θέλετε να βγείτε από την αίθουσα, μπορείτε να εγκαταλείψετε την αίθουσα, αλλά αθόρυβα. Όχι ε, με προκαλώντας ε, θόρυβο. Υπάρχει αρκετός ε, χώρος έξω από την αίθουσα για να συνεχίσετε τις κατηδίαν συζητήσεις. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει η Επιτροπή. Λοιπόν, κύριε Χούτμαν, σε πάρα πολλούς σημαντικούς τομείς η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπόρεσαν να επιτύχουν τους στόχους τους. Εμείς ε, θεωρούμε ότι αν δεν υπάρχει μια στρατηγική για την αστική κινητικότητα, δηλαδή ε, κλιματική αλλαγή, ε, θέματα υγείας, περιφερειακής ανάπτυξης, τεχνολογικής εξέλιξης, αν δεν συνδεθούν όλα αυτά δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Εξάλλου, οι στόχοι της πολιτικής μεταφορών δεν μπορούν να επιτευχθούν αν δεν εξεταστεί το θέμα της ε, αστικής κινητικότητας. Γιατί οι αστικές μεταφορές είναι αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, οι αστικές περιοχές ε, βρίσκονται εν τη γενέση και είναι και στόχος ε, των μεγαλύτερων ροών μεταφοράς που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αφορά βεβαίως και τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Όπως γνωρίζετε, η αστιφιλία είναι μία από τις ε, σημαντικότερες προκλήσεις που επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον των μεταφορών. Αυτό ως ε, έκθεση εγκρίθηκε τον Ιούνιο. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο η ενδιάμεση αναθεώρηση της Λευκής Φίβλου περί μεταφορών που ανακοινώθηκε το 2006 εξετάζει την προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση από τον τομέα της αστικής κινητικότητας. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Πράσινης Βίβλου ε, διαβουλευθήκαμε εκτενώς με τους άμεσα εμπλεκόμενους για να υπάρξει ένας νέος πολιτισμός για την αστική κινητικότητα. Τη στιγμή που αυτό μας έχει βοηθήσει έτσι και αλλιώ να χαράξουμε μια πολιτική ε, νέα δίδοντας σημασία σε διαφορετικούς τομείς. Εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να, ε, το ότι συνέβαλαν οι μεμονωμένοι πολίτες και οι εμπλεκόμενοι, γιατί όλοι αυτοί θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει ρόλο στον τομέα της αστικής κινητικότητας. Τώρα, το πρόγραμμα δράσης εγκρίθηκε στις 30 ε, Σεπτεμβρίου, προτείνει 20 μέσο μακροπρόθεσμα, μάλλον βράχη μεσοπρόθεσμα μέτρα μέχρι το 2012 Πάρα πολλά μέτρα προτείνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη δική του την έκθεση πρωτοβουλίας ε, του Απριλίου και αυτά συμπεριλαμβάνονται και στο τελικό κείμενο της δικής μας, ε, του δικού μας ε, προγράμματος δράσης. Ήδη έχουμε οργανώσει τις δράσεις γύρω από έξι ομάδες που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες που θα προκύπτουν κατά τη διαβούλευση για την πράσινη βίβλο. Οι δράσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και επιπλέον συμπληρώνουν και άλλες πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε άλλους τομείς. Προγραμματίζουμε λοιπόν να έχουμε αναθεώρηση ε, της εφαρμογής του προγράμματος δράσης το 2012 και τότε θα αποφασίσουμε κατά πόσον θα δρομολογήσουμε και άλλες δράσεις σε αυτό τον τομέα. Τώρα, οι έξι αυτές ομάδες είναι οι εξής. Η πρώτη ομάδα αφορά την προαγωγή ολοκληρωμένων πολιτικών ε, με ένα θέμα στόχο που είναι η προαγωγή βιώσιμων προγραμμάτων αστικής κινητικότητας. Αυτό είναι το κλειδί για την ε, βιώσιμη κινητικότητα. Στον τομέα αυτό ε, θα υπάρξει και συσχετισμός με την βιώσιμη κινητικότητα στην ε, περιφερειακή πολιτική και με την υγεία στο περιβάλλον. Το δεύτερο θέμα εστιάζεται στους πολίτες και εντοπίζει τα δικαιώματα των πολιτών στις ε, δημόσιες μεταφορές, βελτιωμένη ε, προσπελασιμότητα για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, καλύτερη ενημέρωση των ταξιδιωτών, πρόσβαση σε πράσινες ζώνες, ε, υποστήριξη εκστρατιών για την κινητικότητα και κάποια πεδία σε θέματα οδήγησης. Το τρίτο θέμα καλύπτει το πρασίνισμα, το πούμε έτσι, των αστικών μεταφορών, που περιλαμβάνει δράσεις για να ενισχυθεί η έρευνα και προγράμματα επίδειξης ε, για ε, αυτοκίνητα με χαμηλές εκπομπές, μία μελέτη για τα αστικά στοιχεία της εσωτερήκευσης του εξωτερικού κόστους και μία μελέτη για την ανταλλαγή πληροφοριών ε, για τα ε, συστήματα κοστολόγησης αστικής κινητικότητας. Το τέταρτο θέμα αφορά τη χρηματοδότηση. Εκεί θέλουμε να ενισχύσουμε την κοινοτική χρηματοδότηση, πρώτα απ' όλα βελτιώνοντας τους υπάρχοντες πόρους, αυτή να είναι περισσότερο διαθέσιμη, να υπάρχει καλύτερο συντονισμός και θέλουμε και να αναλύσουμε την ανάγκη για μελλοντική χρηματοδότηση, έχοντας κατά νου τη νέα δημοσιονομική προοπτική πέμπτο θέμα. Εκεί θα ανταλλάξουμε εμπειρίες και γνώσεις έτσι ώστε να έχουμε δράσεις για να αναβαθμιστούν τα δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία. Θα υπάρξουν δράσεις για τη διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών, έτσι ώστε να υπάρχει ένα παρατηρητήριο. αφού το πήραμε από την έκθεση του Κοινοβουλίου τον Απρίλιο. Και επίσης επιθυμούμε να διευκολύνουμε τον διεθνή διάλογο και την ανταλλαγή πληροφοριών. Και τέλος, το τελευταίο θέμα είναι ότι θα βελτιστοποιήσουμε την αστική κινητικότητα όσον αφορά ε, τις ε, μεταφορές ε, εμπορευμάτων και ευφύ συστήματα μεταφοράς. Το πρόγραμμα δράσης, εμείς δεν περιμένουμε αυτό να δρομολογήσει συγκεκριμένες ενέργειες. Ήδη τους τελευταίους μήνες διοργανώσαμε διάφορες ενέργειες ε, στον τομέα της αστικής ε, κινητικότητας ε, προς τα τέλη Μαρτίου και τώρα πρόκειται να δρομολογήσουμε και τα έξι αυτά επιλεγμένα προγράμματα που σας ανέφερα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει δύο μελέτες. Η μία έχει σχέση με τις πράσινες ζώνες και αξιολογεί την ύπαρξη αλλά και τον προγραμματισμό περιβαλλοντικών ζωνών. Γίνονται ε, προτάσεις ε, για την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Αυτό θα βοηθήσει στο να εντοπιστεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα σε περιβαλλοντικούς και κινητικούς στόχους. Η δεύτερη μελέτη θα εξετάσει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληρωμής ε, και εισιτηρίων στα διάφορα μέσα μεταφοράς. Έχουμε ήδη ανοίξει ένα site στο διαδίκτυο για να βοηθήσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες έτσι ώστε να αγοράσουν ε, καθαρά και αποτελεσματικά μέσα μεταφοράς. Πιο καθαρά λεωφορεία για τις δημόσιες μεταφορές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Χούτμαν. Έχω από την πλευρά της Επιτροπής των Περιφερειών μαζί με τον Αλμπόρο, διότι ζήτησε η Επιτροπή των Περιφερειών να συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση με μεγάλη ευχαρίστηση. Δέχτηκα να γίνει κάτι τέτοιο. Θα δώσω λοιπόν τη δυνατότητα να λάβει το λόγο <clears throat> και πριν από του συντονιστέ μα και πριν από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπράγαν. Συγγνώμη που καθυστέρησα λιγάκι. Ξεκινώ λέγοντα ότι ελπίζω, ελπίζω να μπορέσουμε να προωθήσουμε και τα θέματα που σας ενδιαφέρουν και εσάς και τα θέματα της αστικής κινητικότητας αλλά συγχρόνω και τα θέματα που ενδιαφέρουν τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ, δηλαδή την Επιτροπή των Περιφερειών. Έχουμε συνεργαστεί <clears throat> πολύ στενά με τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκθεση πρωτοβουλία για το θέμα αυτό, τον Αλέν Σαβαρή, με στόχο να αναπτύξουμε όχι μόνο μια δική μα απάντηση <clears throat> για την γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου, αλλά για να μπορέσουμε να διατυπώσουμε και μια δική μας γνωμοδότηση στην Επιτροπή των Περιφερειών έναντι και της έκθεσης του Κοινοβουλίου, που ήταν έκθεση πρωτοβουλία και της ε, Πράσινης Βίβλου της Κομισιόν. Έχει δει, ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Εγώ είμαι εισηγητή από την Επιτροπή των Περιφερειών. Θα συζητηθεί ένα έγγραφο εργασία στην Επιτροπή Εδαφικής Συνεκτικότητας, ΚΟΤΕΡ, στην Επιτροπή των Περιφερειών την επόμενη εβδομάδα. Και ο στόχο μου είναι να έχω το τελικό έγγραφο τον Φεβρουάριο και να το εξετάσει τον Απρίλιο η Ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών. Αυτή είναι λοιπόν μια, ε, ένα χρονοδιάγραμμα που μάλλον θα περατωθεί ταχύτερα από την, το δικό σας χρονοδιάγραμμα. Ελπίζουμε λοιπόν να έχουμε μια στενή συνεργασία με την Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε και η δική μου γνωμοδότηση να περιλαμβάνει ιδέες ε, που θέλετε και εσείς να προωθήσετε και να Εξασφαλίστε θα ληφθούν υπόψη. Τούμπαλιν επίση, νομίζω ότι μπορώ να σας δώσω την απαραίτητη αρρωγή από την πλευρά των τοπικών και περιφερειακών αρχών, ώστε να βοηθήσω το Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα τη δική σα Επιτροπή να διαμορφώσει απόψεις για τα θέματα αυτά. Όπως ελέγχθη, υπάρχει πολύ μικρή διαφορά μεταξύ της Επιτροπής των Περιφερειών και της Κομισιόν σε σχέση με το σχέδιο δράσης έχουν ακούσει τις απόψεις μας, όπως και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολλά από αυτά τα οποία εμείς ζητήσαμε και για τα οποία επιχειρηματολογήσαμε αντανακλώνται στο σχέδιο δράσης. Το πραγματικό πρόβλημα είναι πάντα το θέμα της επικορικότητας. Νομίζω ότι η Κομισιόν το έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς στην έκθεση για το σχέδιο δράσης, γιατί πάντα ήταν ένα δύσκολο πρόβλημα για να μπορέσουμε να πείσουμε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που έχουν ευθύνη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και οι οποίες θεωρούσαν ότι δεν είχε υπάρξει επαρκής διαβούλευση μαζί τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι λοιπόν που το σχέδιο δράσης αντιμετωπίζει και το θέμα αυτό. Υπάρχουν επίση ορισμένοι τομεί για του οποίου θα ήθελα να υπάρχει μεγαλύτερη αναφορά στο σχέδιο δράση. Έκανα μια συνάντηση προηγουμένω στην Γενική Διεύθυνση Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανέφερα ότι θα έπρεπε να υπάρχει ίσως μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα μεταφόρτωσης και αλλαγής τρόπων μεταφοράς και περισσότερη έμφαση στα σχέδια αυτά <clears throat> μέσα στο πλαίσιο της ε, αστικής κινητικότητας. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να προωθήσουμε περισσότερο τα θέματα που μας ενδιαφέρουν για την αστική κινητικότητα και να τα συμπεριλάβουμε και σε άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν θεωρεί ότι μπορεί να προχωρήσει με εργαλεία τα οποία ήδη υφίστανται. Ίσως όμως θα πρέπει να κοιτάξουμε και πάλι να δούμε αν χρειαζόμαστε νέα εργαλεία και περισσότερο νέα χρηματοδοτικά μέσα για να προωθήσουμε αυτά τα θέματα. Υπάρχουν προβλήματα αστικής κινητικότητας σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων. Ελπίζω ότι αυτή η συζήτηση θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά τα οποία υπάρχουν σε πολλές από τις αστικές περιοχές, σε στα περισσότερα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σερ Άλμπερτ. Ελπίζω να διαβιβάσετε τις ευχές μας, τους χαιρετισμούς μας στην Επιτροπή των Περιφερειών. Κύριος Γκρός. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω και την Κομισιόν για την παρουσίαση της πρότασής της και θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής των περιφερειών και είχαμε ήδη την ευκαιρία να συζητήσουμε για το θέμα αυτό μαζί του στο παρελθόν, γιατί αυτό το θέμα της αστικής κινητικότητας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Δυστυχώς, η επικουρικότητα μερικές φορές χρησιμοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σαν μια τροχοπέδη στις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι η καλύτερη χρήση της επικουρικότητας. Δεύτερη παρατήρηση, έχω διαπιστώσει ότι αν δεν δίνονται χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλα αυτά θέλει να νομοθετεί, όλα αυτά μένουν στο επίπεδο της φιλολογίας, δεν οδηγούν σε συγκεκριμένες δράσεις. Αν δεν υπάρξει σαφή στοχοθεσία λοιπόν, Μπορούμε να συζητήσουμε πώς θα τα εφαρμόσουμε όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν σαφή στόχη και σαφή μέσα για την υποστήριξή του σε χρηματοοικονομικό επίπεδο. Αλλιώς μπορούμε να κάνουμε μελέτες και συζητήσεις ατέρμονες, αλλά δεν θα προχωρήσουμε καθόλου. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια συγκεκριμένη υποστήριξη για την επίτευξη αυτών των στόχων. Επομένω, για αυτό το λόγο πιστεύω ότι όχι μόνο η Επιτροπή των Περιφερειών, αλλά και η δική μα Περιφερειακή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντικοί εταίροι, οι οποίοι θα μπορούσαν να μα βοηθήσουν να έχουμε μια καλύτερη κατεύθυνση των διαρθρωτικών πόρων για τομεί που είναι πραγματικά σημαντικοί τομεί για την περιφερειακή πολιτική. Και επομένω οι πόροι αυτοί οι οποίοι υπάρχουν μέσα στη διαρθρωτική πολιτική, όπως και να ότι, ότι οποιοδήποτε τίτλο και να έχουν πάνω το κεφάλι τους θα πρέπει να μας βοηθήσουν να βοηθήσουμε την αστική κινητικότητα. Παραδείγματο χάρη θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ποσά τα οποία αποκτούμε από τη χρήση της Ευρωβινιέτας για την ε, προώθηση της αστικής κινητικότητας. Θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν να πάρουμε τέτοιες πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε να συνδέσουμε την αστική κινητικότητα στα κρατημέλη μας με μια ευρύτερη συζήτηση. Μια ακόμα παρατήρηση Πιστεύω ότι θα πρέπει η επικουρικότητα να μην εμποδίσει την ανάπτυξη μιας πραγματικής συνεκτικότητος στις μεταφορές και αυτό αφορά και την μεταφορά από ένα τομέα, από ένα τρόπο μεταφορές σε ένα άλλο τρόπο μεταφοράς. Και στο συγκεκριμένο αυτό έγγραφο θα πρέπει να παραμείνουν όλα αυτά μέσα σε ένα συνεκτικό πλαίσιο. Αυτά λοιπόν τα οποία καθορίζονται σαν στόχοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο με διαφορετικό τρόπο. Για μένα λοιπόν το σημαντικό είναι υποστηρίζω την ε, επικουρικότητα αλλά όχι σαν πρόσχημα για να μην γίνει τίποτα. Δεύτερον θα πρέπει να υπάρχει μια προσπάθεια συγκεκριμένου στόχους και συγκεκριμένη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων με παλιά ή και νέα μέσα. Και τρίτον, να εξασφαλίσουμε τη συνεκτικότητα των δράσεών μα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή ενώπιόν μας ως σχέδιο δράσης, πιστεύω ότι σε ορισμένου τομεί είναι πράγματι πλήρες, σε άλλους τομείς είναι λιγότερο πλήρες. Αυτό το οποίο εμένα με ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση είναι ποια θα είναι τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα με τα οποία θα εφαρμόσουμε στην πράξη όλα αυτά, ώστε να μην μείνουν σε ένα ακαδημαϊκό επίπεδο, να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα για το ποιο στόχο θα επιτευχθεί σε ποιο χρονικό ορίζοντα Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συνεργαστούμε και με την Επιτροπή των Περιφερειών και ελπίζω και σε άλλους τομείς θα μπορέσουμε να εργαστούμε ώστε τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες της Ευρώπης να είναι εταίροι στη χάραξη πολιτικής. Πιστεύω λοιπόν ότι η εμβάθυνση της σχέσης μας, και αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, ένα πολύ καλό παράδειγμα, θα ήταν χρήσιμο να μην χάσουμε την ύπαρξη της Επιτροπής των Περιφερειών από τα όματά μας και το ρόλο που μπορεί να παίξει και επίσης να έχει και τα απαραίτητα μέσα για να συνεχίσει το ρόλο της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Αλκαντράουι. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ε, εκπρόσωπο της Επιτροπής των Περιφερειών. Δεν θα επαναλάβω τώρα γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σχέδιο δράσης πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Τακτικά το συζητήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια το θέμα και χαίρομαι που υπάρχει ένα σχέδιο δράσης και επιπλέον σε μεγάλο βαθμό έχει λάβει υπόψη τις προτάσεις μας, τις προτάσεις του συναδέλφου μου, του κυρίου Σαβαρή και άλλων. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέφθασε αργότερα από ό,τι περιμέναμε. Τα είχαν υποσχεθεί ότι θα πούν κάτι το τέλος του περασμένου έτους, ας το ξεχάσουμε. Τώρα το σχέδιο και το πόσο αποτελεσματικό θα είναι εξαρτάται από το κατά πόσο θα τηρήσει τις ε, υποσχέσεις της η Επιτροπή. Υπάρχει ένας κατάλογος προτάσεων, ε, μια φετηρία για κάθε πρόταση, χρονική. Πολύ συχνά όμως δεν περιγράφονται πολλές λεπτομέρειες και δεν ποσοτικοποιούνται τα στοιχεία. Όπως και ο κύριος Γκρός και εγώ θα πω ότι ελπίζω να έχουμε κάποιους σαφείς στόχους, πρακτικούς στόχους και κάποιες προθεσμίες που θα αναφέρονται. Και έτσι θα μπορέσουμε να μπούμε στις πρακτικές λεπτομέρειες της προσπάθειας. Από την πλευρά μου, όσον αφορά την πρώτη φάση, νομίζω ότι προτεραιότητα θα πρέπει να δώσουμε στην ανάπτυξη ενός καλού συστήματος ανταλλαγής ιδεών. Υπάρχουν πολλές πόλεις που ε, διενεργούν, εφαρμόζουν μάλλον πιλωτικά προγράμματα, δοκιμαστικά προγράμματα και προσπαθούν να βελτιώσουν την κινητικότητα και να την κάνουν πιο βιώσιμη. Για να πετύχουμε αυτό το στόχο, κάτι που αναφέρεται και στο σχέδιο δράσεως, χρειαζόμαστε αξιόπιστες πληροφορίες, καλές πληροφορίες. Το συζητήσαμε αυτό την περασμένη φορά στην Επιτροπή μας. Χρειαζόμαστε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία αξιόπιστα δεδομένα που θα πρέπει να συλλέγονται, ούτως ώστε να γίνεται η σωστή σύγκριση και να μπορέσουμε να κάνουμε ανάλυση ε, συνεπιών πιο ορθή. Υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα σχετική ιδέα που αναφέραμε όσον αφορά τη δημιουργία μιας Επιτροπής Ελέγχου για την Κινητικότητα, ένα είδος παρατηρητηρίου. Αναφέρεται σε ένα εικονικό δίκτυο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αρχική φάση. Συμφωνώ ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα χωρίς να δημιουργηθεί άλλη, άλλη μια στιβάδα γραφειοκρατική, ένα εικονικό δίκτυο θα μπορούσε να είναι κάτι καλό, αλλά να δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι πόλεις να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Να είναι εύκολο να το χρησιμοποιήσουν το δίκτυο αυτό και να βρουν πληροφορίες. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να γίνει μια εκστρατεία ενημέρωσης της πόλης, να μάθουν στις πόλεις ότι υπάρχει αυτό το εργαλείο, ότι μπορεί να τους βοηθήσει, ούτως ώστε να δώσουν καλές ιδέες και να μάθουν οι διάφορες πόλεις από τις εμπειρίες άλλων πόλεων. Θα ήθελα να ακούσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει πώς το βλέπει το θέμα, πώς προτίθεται να, προτίθεται να το ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πρέπει να ξεκινήσει όλη η προσπάθεια φέτος. Άλλη σειρά μέτρων αφορά τη χρηματοδότηση και την ενθάρρυνση της εισαγωγής νέων τεχνολογιών αυτό είναι ένα δεύτερο σημαντικό θέμα κατά την άποψή μου, όπου εκεί μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία η Ευρώπη. Όσον αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης, όπως είπα υπάρχουν πολλές ε, δυνατότητες, θα πρέπει κάπως να συντονιστούμε και να επιβάλλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και να είναι πιο ορατή η χρηματοδότηση στις πόλεις, πού μπορούν να αποτανθούν για να πάρουν χρήματα, ποιες δυνατότητες υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για χρηματοδότηση η κινητικότητα θα πρέπει να έχει μεγάλη προτεραιότητα, κατά την άποψή μου, όταν συζητούμε τις επόμενες δημοσιονομικές προπτικές, επί παραδείγματι, θα πρέπει να είμαστε πιο δραστηροί και να προσπαθήσουμε όλα αυτά να τα προβάλλουμε περισσότερο. Να έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στον επόμενο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσης όσον αφορά την έρευνα, τυποποίηση, νέα τεχνολογία και εκεί θα πρέπει να έχουμε ένα σφαιρικό όραμα και να συνεργαστούμε να συνεργαστούν οι Γενικές Διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το σκοπό. Αυτές λοιπόν είναι οι βασικές προτεραιότητες. Προφανώς υπάρχουν κι άλλες και θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει ε, ποια συνέχεια θα δοθεί στο σχέδιο δράσεως. Αναφερθήκατε στο 2012 σαν ε, χρονολογία για την αποτίμηση, για την αξιολόγηση και κατά πόσο θα, θα χρειαστεί ένα νέο σχέδιο δράσης βάσει της αποτιμήσεως. Το ερώτημα είναι το εξή. Βάσει του ισχύοντος σχεδίου δράσεως, Μπορεί να μας δώσετε λεπτομέρειες. Τι θα κάνετε φέτος, του χρόνου, το 2011, πιο πολλές λεπτομέρειες. Πώς θα μας ενημερώνετε όσον αφορά την πρόοδο των μέτρων αυτών, το πώς θα εφαρμόζονται. Υποτίθεται ότι ξεκινάτε το 2009, ότι ξεκινάει κάτι το 2009 και άλλα εφαρμόζονται το 2010. Πότε θα υλοποιηθούν όλα αυτά. Αυτό είναι σημαντικό να το ξέρω. Παραδείγματο χάρη, μπορούμε να συμφωνήσουμε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο, θα έρχεστε εδώ στην Επιτροπή μας να μας ενημερώνετε σχετικά με τις εξελίξεις πού βρίσκονται τα διάφορα μέτρα που έχετε δρομολογήσει, ούτως ώστε εμείς εδώ στην Επιτροπή να έχουμε μια γενική εικόνα των όσων συμβαίνουν. Η κυρία Μάισνα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά ε, την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλες τις πολιτικές ομάδες να ευχαριστήσω και την Επιτροπή των Περιφερειών για όλα αυτά που μας είπατε. Νομίζω ότι μπορώ να συνεχίσω ακριβώς εκεί που το άφησε η προλαλή σας. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό το ότι στο πρόγραμμα δράσης έχουμε συγκεκριμένες ε, προτάσεις οι οποίες πραγματικά μπορούν να συμβάλλουν στο να προαχθεί περαιτέρω η αστική κινητικότητα. Με αυτό το πρόγραμμα δράσης. Εξάλλου αυτός είναι και ο στόχος μας. Και εδώ επιτρέψτε μου να προσθέσω ορισμένα στοιχεία Πρώτον, η βιώσιμη κινητικότητα, αυτή που είναι διαρκείας, που κατά κανόνα συνδέεται και με ε, μια στάση φιλική προς το περιβάλλον. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Νομίζω το σύνολο της πολιτικής μεταφορών τώρα πλέον θα πρέπει να διαμορφώνεται κάτω από το πρίσμα του περιβάλλοντος και της υγείας. Για μένα λοιπόν όσον αφορά τη διάρκεια πρέπει κανείς να έχει κατά νου πώς αλλάζει η κοινωνία και πώς αλλάζουν και οι απαιτήσει των ανθρώπων για την αστική κινητικότητα. Γιατί αυτή δεν είναι μόνο η προϋπόθεση για μια εύρυθμη λειτουργία της κοινή αγοράς, αλλά είναι και ένα σύνεκουανόν έτσι ώστε η ζωή των ανθρώπων να μπορεί να έχει κάποια ποιότητα. Άλλαξε λοιπόν η κοινωνία. Τώρα πλέον έχουμε περισσότερους ε, υπερήλικες, έχουμε περισσότερους ανθρώπους με περιορισμένη κινητικότητα. Ως εκ τούτου λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και αυτό το επισημάνατε στην έκθεση Κομισιόν ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για το τι μπορεί να βελτιωθεί στις αστικές μεταφορές, κυρίως με άτομα περιορισμένης κινητικότητας. Νομίζω ότι εδώ ε, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα. Δηλαδή, οι άνθρωποι με αναπηρία πώς μπορούν να αποκτήσουν τις πληροφορίες γιατί εδώ ας πούμε, ε, θα μπορούσαν να υπάρχουν ειδικοί πίνακες ε, με ειδικό φωτισμό ή ε, με γραφή μπρέι. Αυτά είναι συγκεκριμένα παραδείγματα και νομίζω με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να περάσει στην ουσία της βιώσιμης κινητικότητας. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό για μένα και δεν, τέθη, δεν, αναφέρθηκε εδώ στις προφορικές παρεμβάσεις, παρότι περιλαμβάνεται ε, στην έκθεση. Πρόκειται για την ITS. Υπάρχει ο στόχος που είναι να περιοριστεί ο αριθμός ε, των ε, θυμάτων από τροχαία ατυχήματα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα στατιστικά δεδομένα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι μοντέλα όπως open space, ανοιχτός χώρος, που έχει δοκιμαστεί το μοντέλο αυτό. Εντάξει, δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις πόλεις, αλλά έχει εφαρμοστεί. Και είδαμε ότι με τέτοια μοντέλα ε, τέτοια μοντέλα βελτιώνουν την ασφάλεια και δεν ε, παρεμποδίζουν την λειτουργία Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά είναι σημαντικά και εμένα θα με ενδιαφέρει να μάθω να ψήφω αυτά. Ευχαριστώ κυρία Λεκτεμπέργα. Ευχαριστώ πολύ. Η πρόταση για τον ανοιχτό χώρο, την χρήση του ακάλυπτου χώρου, δηλαδή ίσως θα έπρεπε να το δοκιμάσουμε και στις Βρυξέλλες. Για μένα το, ένα από τα ουσιαστικά ερωτήματα σε όλη αυτή την προβληματική είναι πάντα όπως ανεφέρθηκε προηγουμένως το θέμα της επικουρικότητας. η οποία θα πρέπει να γίνεται με ένα θετικό τρόπο η εφαρμογή της επικουρικότητας. Γιατί ορισμένοι λένε ότι είναι πολύ προχωρημένοι, ενώ άλλοι ίσως υπολείπονται στα θέματα αυτά της αστικής κινητικότητας και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά εμπόδια. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα έτσι ώστε οι προχωρημένοι, οι οποίοι είναι καινοτόμοι, να μην τροχοπεδούνται και συγχρόνως αυτοί οι οποίοι υπολείπονται να έχουν τα κατάλληλα κίνητρα για να πράξουν τα απαραίτητα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πραγματικό, το ουσιαστικό ερώτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για τις προτάσεις τις οποίες έχει θέσει, αλλά χωρίς συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένα χρονοδιάγραμματα, φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει σε ακινησία και, μη έλλειψη, και έλλειψη δράσης. Νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε σε στόχο να έχουν όλοι οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη την δυνατότητα να απολαμβάνουν τη αστική κινητικότητα και όχι μόνο αυτοί που ζουν σε κράτη τα οποία έχουν ήδη αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό με ένα επωφελή τρόπο. Πώ λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα για μένα, πώ θα καταφέρω παρά την επικουρικότητα ή ακόμα και χάρη στην επικουρικότητα να καταλήξω στα κατάλληλα αυτά μέτρα τα οποία θα εξασφαλίσουν να υπάρχει ενεργή δράση από όλους και θα ήθελα ακριβώ να ξέρω ποια είναι η αντιμετώπιση, η αντίληψη που έχει η Κομισιόν για να λύσει αυτό το πρόβλημα, γιατί σε, από αυτό εξαρτάται η πρόοδος. Δεν αρκεί να θέτουμε στο διαδίκτυο τις ε, βέλτιστες πρακτικές και τις ε, προτάσεις, γιατί μπορεί το κάθε κράτος να πει ότι στη δική μου περίπτωση, στις συγκεκριμένες μου πόλες, αυτό το σύστημα το οποίο είναι τόσο έξυπνο και καινοτόμο δεν θα λειτουργήσει. Αν δεν υπάρχει λοιπόν η πίεση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα η κάθε χώρα με την πίεση των πολιτών της δεν θα επιτευχθεί τίποτα. Πώς λοιπόν αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα εσείς, πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και για μένα είναι ένα από τα κεντρικά ερωτήματα. Χωρίς να έχουμε συγκεκριμένους στόχους με πληθώρα μεθόδων και προτάσεων δεν μπορούμε πραγματικά να καταλήξουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το 2012 θα έχουμε πράγματι πραγματοποιήσει κάτι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στις μεταφορές είναι ότι δεν έχουμε αρκετή φιλοδοξία η οποία να εκφράζεται από την πλευρά των κρατών μελών. Κύριε Απόστα. Yeah, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρον το έγγραφο. κάνει τα πάντα, θέλει να κάνει τα πάντα και αυτό είναι μη ρεαλιστικό θα έλεγα. Το διάβαζα. Και πολλά στοιχεία του περιεχομένου αφορούν πράγματα που συζητούσαμε στην Επιτροπή εδώ και δέκα χρόνια. Αστική κινητικότητα κλπ. Είναι θέμα επικουρικότητας. Εγώ δεν είμαι αντίθετη στη συνεργασία, βεβαίως. Έχουμε περιφερειακές επίτροπες και ξέρουμε ότι συνεδριάζουν και εξετάζουν τις βέλτιστες πρακτικές και προσπαθούν να δουν τι ισχύει σε μία πόλη, τι ισχύει σε μία άλλη πόλη. Δεν ε, καταλαβαίνω τι θέλουμε να κάνουμε. Είναι πολύ παλιά τα επιχειρήματα που συμπεριλαμβάνονται. Διαβάζω στο κείμενο, χωρίς να θέλω να είμαι σκληρή, πρέπει να πω ότι εκπλήσω με τα μάλα από κάποια σχόλια. Συνεργασία, ναι, πάση θυσία βεβαίω. Το διαβάζουμε το κείμενο και την μια πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διατείνεται τον θέμα επικουρικότητας και το αναγνωρίζει και το επόμενο ε, που κάνει είναι να μειγνύεται στα πάντα ή θα να θέλει να αναμειχθεί. Προσφέρει εταιρικέ σχέσει. Πολύ καλό αυτό. Εγώ δεν έχω πρόβλημα τι εταιρικέ σχέσει. Αλλά πού ταιριάζει αυτό, τι σημαίνει. Στο πρώτο θέμα, στη σελίδα 4, Ολοκληρωμένη προσέγγιση δεν είναι κάτι που απαιτείται μόνο για την ανάπτυξη υποδομών, μεταφορών κλπ. Το ξέρουμε αυτό. Αυτό κάνουμε, αυτό μιλάμε, αυτό συζητάμε. Αυτό συζητά η τοπική αυτοδίκηση. Τι πράγμα συζητούμε, διότι αυτό αφορά την τοπική αυτοδίκηση, εθνικές κυβερνήσεις κλπ. Στη σελίδα 5, σχέδιο δράσεως 3, εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών, το συζητάμε. Και λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει, και το λέω σοβαρά αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων προ υγιεινό περιβάλλον και θα διερευνήσει στα πλαίσια των εργασιών τη όσον αφορά τη δημόσια υγεία, κυρίω την εφαρμογή στρατηγικών όσον αφορά τη διατροφή, ε, παχυσαρκία, περιβάλλον, υγεία, πρόληψη καρκίνου, τραυματισμών κλπ. Δεν καταλαβαίνω, ανησυχώ τα μάρα, τι διαβάζω εδώ. Διαβάζω ένα έγγραφο που εξετάζει τα θέματα κινητικής, ε, αστικής κινητικότητας. Προσπαθούμε να πάμε το σημείο α στο σημείο β. Αυτό είναι πρόβλημα για τους ανθρώπους που ζουν στην πόλη και πώς αυτά ταιριάζουν με αυτό το πλαίσιο. Δεν είμαι σίγουρη. Και κάτι άλλο. Μ' ανησυχούν αυτά που σας ε, θίγω. Είναι καλό να συζητάμε καλά τα βήματα που θα κάνουμε για να προχωρήσουμε σε διάφορους τομείς. Για την κοστολόγηση. Κάτι φοβερό είδα, σελίδα 7. Ρυθμιστική Επιτροπή για άδειε οδήγηση. Μπορούμε να σας πούμε δηλαδή πώς να οδηγήσετε για να μην χρησιμοποιείτε πολλά καύσιμα. Αυτό μυρίζει έτσι από... Ε, σαν να έχεις τη μαμά, την κουβερνάντα πάνω το κεφάλι σου. Ε, μπορεί να συζητά κανείς την επικουρικότητα, να συζητά κανείς το θέμα της συνεργασίας, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ο στόχος ή οι στοχη Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε. Ξέρουμε τι θέλουμε να δούμε. Αλλά το έγγραφο, τι είναι αυτό. Σχέδιο δράσης. Άρα έχουμε σχέδιο δράσης. Όλα για όλους, τα πάντα για τους πάντες. Όσον αφορά την Επιτροπή Μεταφορών. Τι συζητάμε. Τι μας αφορά, τι αφορά το δικό μας ρόλο στην Επιτροπή Μεταφορών που δεν κάνουμε, που θα μπορούσαμε να κάνουμε και που δεν συμπεριλαμβάνεται σε κάποιο σχέδιο οδηγίας, ITS ή μεταφορά εμπορευμάτων. Έχουμε οδηγίες, έχουμε προτάσεις που εξετάζουν κάποια αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, εγώ εδώ πέρα βαδίζω στα σκοτεινά. Εγώ δεν τα έθεσα ως αστεία αυτά, δεν νομίζω την αστεία αυτά τα σημεία. Τα έθεσα γιατί είμαι περίεργη, δεν καταλαβαίνω περί τίνος πρόκειται. Τι ακριβώς στόχο έχει αυτό το έγγραφο. Ο Αντιπρόεδρος Μαντάλεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το θέμα της επικορικότητας είναι κομβικό θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά από αυτά που είπε η κυρία Φώστερ Αυτά είναι θέματα τα οποία θα συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια. Όχι μόνο δέκα χρόνια όπως ελέγχθη. Ήδη από το τέλος της δεκαετίας των 1980 είχαμε αρχίσει να συζητάμε για αυτό το θέμα και την σύνδεσή του με την επικορικότητα. Πιστεύω <clears throat> ότι εδώ θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να κάνουμε την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και να έχουμε μια πλατφόρμα που θα μας επιτρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο, παραδείγματος χάρη μέσω του διαδικτύου. Εγώ δεν ανησυχώ με αυτά που ανέφερε η κυρία Λίχτεμπεργκ, γιατί πάντα στα κράτη-μέλη υπάρχουν άτομα με μεγάλη ικανότητα και επομένως αν μέσα από αυτή την πλατφόρμα ανταλλαγής βελτίστων πρακτικών μπορούν να αποκτήσουν ιδέες για το τι μπορούν να κάνουν σε τοπικό επίπεδο, πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε λοιπόν πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αντιμετωπίζει. Καταρχήν η Ευρώπη δεν έχει προβλήματα όπω αυτά τα οποία έχουμε πόλει, όπω το Σαν Φρανσίσκο που ανεβαίνει κανεί και μετά ξεχνάει να κατέβει. Τέτοιου δρόμου που είναι πάρα πολύ δύσκολου Εγώ ω Ολλανδό υποστηρίζω ιδιαίτερα το να χρησιμοποιούμε στο βαθμό του δυνατού τα ποδήλατα και στι πόλει. Έχουμε πολλά παραδείγματα τα οποία μας καταδεικνύουν ότι ο καλύτερος, ο ταχύτερος τρόπος μετακίνησης σε μία πόλη είναι το ποδήλατο. Οποιαδήποτε πόλη λοιπόν <clears throat> θέλει να επωφεληθεί από τις εμπειρίες μας, είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε τα στοιχεία αυτά. Η επικουρικότητα λοιπόν είναι πολύ καλή, αλλά και η ανταλλαγή απόψεων είναι πάρα πολύ θετική και εμείς είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε τα δικά μας στοιχεία. Θέλετε να απαντήσετε. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορώ ακόμα να πάρω το λόγο. να μιλήσω. Ε, μισό λεπτό την κυρία Γιαναλόβα. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε. Δεν άκουσα καλά το όνομά μου. Εγώ θα ήθελα να μοιραστώ τις εμπειρίες μου. Προέρχομαι από μια πόλη που συμμετέχει εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας της Κινητικότητας που θεωρώ σαν προσπάθειες μεμονωμένες απλώς κάποιων πόλεων δυστυχώς. Τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε το περιβάλλον των πόλεων. Πώς μπορούμε να κάνουμε πιο δραστήριες ε, της πόλης. Ε, ευχαριστιέμαι διότι βλέπω ότι γίνονται καλές προσπάθειες από πλευράς πόλεων στο σχέδιο δράσης, αλλά δυστυχώς είναι τέτοια η πραγματικότητα και έτσι δημιουργούνται νησίδες. Οι πόλεις αποτελούν μεμονωμένες νησίδες που καταβάλουν προσπάθειες. Και πρέπει να υπάρχει γενικότερη προσπάθεια Υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που πάνε κατά της αυξήσεως της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στα νέα κράτη-μέλη. Βέβαια, είναι μια πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε λόγω ανάπτυξη, όπως και η διάλυση των κρατικών, των δημόσιων μέτρων μεταφοράς. Χωρίς χρήματα δεν γίνεται τίποτα. Όταν μιλήσαμε για στόχους σαφείς και προθεσμίες, είναι σωστό να υπάρχουν και τα μέσα για να κινητοποιηθούν οι θετικές δραστηριότητες. Χρειάζονται χρήματα για τη δημιουργία υποδομών, πολύ σημαντικό αυτό, διότι σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά τις υποδομές και εγώ υποστηρίζω ένθερμα την ενίσχυση των μέσων χρηματοδότησης για την τόνωση των υποδομών, για την ποδηλασία, για τα μέσα μαζικών μεταφορών, όλες τις εναλλακτικές μορφές μεταφορών, εναλλακτικέ όσον αφορά τη χρήση των ΙΟΤΑΧΗ. Αυτά και ευχαριστώ. Η κυρία Χούτμαν έχει το λόγο. Τώρα είναι η σειρά σας, πραγματικά είναι η σειρά σας κυρία Χούτμαν. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή να ανταλλάξουμε απόψεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι είναι σαφές ότι η Κομισιόν όπως και στο παρελθόν είναι πάντα έτοιμη μια-δυο φορές το χρόνο να σας δίνει εκθέσεις για την πρόοδο που έχουμε επιτύχει σε σχέση με αυτό το σχέδιο δράσης. Δεύτερον, χαίρομαι που ο κ. Κατρόη έχει αναφέρει και το θέμα της συνεργασίας με άλλες γενικές διευθύνσεις, γιατί πράγματι είναι αυτό ένα θέμα το οποίο και στη φάση προετοιμασίας και στη φάση της ε, υλοποίησης απαιτεί τη συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες της Κομισιόν και πριν να ήταν και μεγάλη ευχαρίστηση για μας. Εργαστήκαμε πολλά άτομα στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης γιατί έχουν μεγάλη πήρα στον τομέα της χρήσης των κοινωνικών πόρων, των διαρθρωτικών μάλλον πόρων και σε όλα τα θέματα της ε, κινητικότητος και της αστικής ανάπτυξης. Εργαστήκαμε με πολλούς συναδέλφους επίσης για θέματα υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας, για τα εφία συστήματα κινητικότητος με τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών κτλ. Και οικοθενοείται και με τους συναδέλφους από την Γενική Διεύθυνση Έρευνα και Ανάπτυξης, διότι χρησιμοποιούμε και την χρηματοδότηση του προγράμματος πλαισίου. Σε σχέση τώρα με το θέμα της επικουρικότητας, η οποία αναφέρθηκε κατά κόγον. Θέλω να διευκρινίσω ότι η επικουρικότητα δεν σημαίνει ότι η Κομισιόν ή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να κάνουν τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι το κατάλληλο εργαλείο σε αυτό το τομέα, γιατί φυσικά είναι οι τοπικές αρχές οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα τα τεκτενόμενα στις πόλεις και στους δήμους, το κατάλληλο εργαλείο είναι η παροχή κινήτρων. Αυτό το οποίο η Κομισιό θέλει να κάνει να ενθαρρύνει τις πόλεις να δράσουν <clears throat> προς την κατεύθυνση της εφαρμογής γενικών πολιτικών που θα ευνοήσουν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα υποστηρίξουν την υγεία, θα αντιμετωπίσουν τη συμφόρηση, θα βελτιώσουν λοιπόν την αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών και επίσης με τον τρόπο αυτό να ενισχύσουμε αυτούς οι οποίοι θέλουν να δράσουν μέσω παροχής πληροφοριών, μέσω χρηματοδότησης, παροχής ε, στοιχείων, ανταλλαγής βελτίστων πρακτικών. Όλα αυτά λοιπόν τα εργαλεία τα οποία εμείς έχουμε αναφέρει στα πλαίσια του σχεδίου δράσης. Εγώ εκπλήσω όταν μου λέτε ότι οι δράσει μας δεν είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένες. Μπορεί να μην είναι λεπτομεριακέ, αλλά όπω ξέρετε η Κομισιόν έχει ένα όριο σε 22.500 αλφοαριθμητικούς χαρακτήρες όταν διατυπώνει τις προτάσεις της. Έχουμε λοιπόν κατά κάποιο τρόπο ζουληχθεί μέσα σε αυτό το πολύ στενό χώρο σε ό,τι αφορά τις προτάσεις μας, αλλά είμαστε πάντα έτοιμοι να σας δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες σε όσους θέλουν. Μερικές από τις παρεμβάσεις των βουλευτών ανέφεραν ότι είναι παλιά τα επιχειρήματα τα οποία αναφέρουν και δεν υπάρχει τίποτα το κενό, το φανές. Δεν είναι πρώτη φορά που η Κομισιόν δράει για τα θέματα αυτά. Εμείς έχουμε αντιμετωπίσει την αστική κινητικότητα σαν τμήμα των πολιτικών μας από το 1995. Δεν είναι απόλυτα λοιπόν νεοφανή όλα αυτά. Αυτό το οποίο είναι καινούριο είναι ότι για πρώτη φορά σε ένα συνεκτικό πλαίσιο θέτουμε όλες αυτές τις δράσεις που είχαμε στο παρελθόν και τις οποίες θα εξακολουθήσουμε να εφαρμόσουμε και στο μέλλον. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ σημαντική άσκηση να έχουμε ένα τέτοιο πλαίσιο συνεκτικό και αυτή την... το σύνολο αυτών των πολιτικών που αφορούν αυτό το τομέα. Λυπάμαι τώρα αν υπάρχουν προβλήματα κατανόησης μου δημιουργούν εντύπωση που δεν κατανοείται το αγγλικό κείμενο, το οποίο είναι και η αρχική μορφή της πρότασης της Κομισιόν. Θα έπρεπε να είναι σαφέστερο από το κείμενο στα αγγλικά, αλλά θέλω να ζητήσω συγγνώμη και από αυτούς οι οποίοι ε, είναι αναγνώστες σε άλλες γλώσσες. Ξέρω ότι δεν έχουν ακόμα αναθεωρηθεί όλες οι μεταφράσεις και γι' αυτό δεν μπορέσαμε να καλύψουμε <clears throat> όλες τις γλώσσες και να εξαλείψουμε τα προβλήματα αυτά. Το αγγλικό κείμενο όμως νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κατανοητό, διότι είναι και το αρχικό κείμενο στο οποίο συντάχθηκε η πρόταση της Κομισιόν. <clears throat> Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αναλλακτικές μεθόδους μεταφορών, όπως είναι η χρήση ποδηλάτων, παραδείγματος χάρη κτλ. Εδώ θέλω να σας αναφέρω ότι τρία από τα σχέδια τα οποία έχω ε, αναφέρει στην πρότασή μου αφορούν απόλυτα την χρήση ποδηλάτων και την πεζοπορία ή αφορούν την χρήση ποδηλάτων σε συνδυασμό με δημόσιες συγκοινωνίες. Όλα αυτά λοιπόν είναι τμήματα των προτεραιοτήτων μας. Υπήρξε και ένα ερώτημα σε σχέση με τα άτομα μειωμένης κινητικότητος και εδώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της κυρίας Μίσνα για την δράση υπαριθμών 5 και να την διαβεβαιώσω ότι η πληροφόρηση σε σχέση με τις ε, μετακινήσεις θα είναι διαθέσιμη και για τους τυφλούς, όπως αναφέρεται στην δράση υπαριθμών 6. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Χούτμαν. Δύο φορές ήρθατε, λοιπόν, παρουσιαστήκατε και μιλήσατε σήμερα. Βγάλετε το ψωμί σα για σήμερα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την, ε, το θέμα αυτό της, της Επιτροπής. Μάλλον στις 5 και 4 το έχουμε συντονιστές. Τελειώσαμε τα σημεία της Επιτροπής. Διακόπτουμε μέχρι τις 5 και 4 για τις συνεδρίες των συντονιστών. Ευχαριστώ τον Σερ Άλμπερτ που ήρθε εκ μέρους της Επιτροπής των Περιφερειών και συντονιστές στις 5 και 4.